Dear colleague, imagine that we can start now. If you can... Uh, Συνάδελφοι, αν ε, θέλετε να καθίσετε για να ξεκινήσουμε, λέει ο Πρόεδρος. Γιατί έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας κάποιους ε, προσκεκλημένους από διάφορα σημαντικά πανεπιστήμια της Ευρώπης. και πολύ χαίρομαι που τους έχουμε εδώ μαζί μας ε, το απόγευμα. Θα σας τους ε, παρουσιάσω. Πέντε καθηγητές και Πριτάνης σημαντικών, όπως έλεγα, πανεπιστημίων. Πανεπιστημίων, με συγχωρείτε, θα συνεχίσω στα Ιταλικά, λέει ο Πρόεδρος. Οπότε φορέστε τα ακουστικά σας. Και φυσικά όλοι μπορούν να μιλήσουν τη γλώσσα τους ή εν πάση εκτός σε όποια γλώσσα επιθυμείτε. Λοιπόν, σήμερα το απόγευμα λοιπόν έχουμε μια ακρόαση ιδιαίτερη σημασία. και να ευχαριστήσω και την Επιτροπή Πολιτιστικών Θεμάτων που ανταποκρίθηκε στην ε, πρόσκλησή μου γιατί νομίζω ότι εντός του πεδίου των αρμοδιοτήτων μας θα πρέπει να συζητούμε ευθέως πιο άμεσα δηλαδή, με τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια αφενός, διότι όπως γνωρίζετε είμαστε απόλυτα δεσμευμένοι στην ενίσχυση των διαφόρων ποιοτικών συστημάτων των, των πανεπιστημιακών φορέων και φορέων ανωτά της εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε και την έκθεση της Κομισιόν, έχουμε την ε, συνάδελφο Λιμπάτσκα που ε, υπέβαλε μια πολύ σημαντική γνωμοδότηση για την διαδικασία της Μπολόνια. Έχουμε την κυρία Σφεντρόβα ε, σχετικά με τις ε, πρωτοβουλίες της υπαχειρηματικότητας. Αλλά πάνω απ' όλα έχουμε το πρόγραμμα Erasmus Plus, το οποίο συμπεριλαμβάνει διάφορες δράσεις, αυτά που ονομάζονται συμμαχίες ή εμπάσχετος εταιρικές σχέσεις της γνώσης μαζί με πανεπιστημιακούς φορείς, οικονομικούς φορείς και επιχειρηματικούς. Μας ενδιαφέρει λοιπόν η άποψή σας σχετικά με αυτό που θα μπορούσε να αντιπροσωπεύει την βελτίωση, την ενίσχυση, τη συμπλήρωση των προγραμμάτων αυτών, των υφισταμένων, του ορίζοντα 2020, του Εράσμους. Είναι ενδιαφέρον αυτό το θέμα και για την Επιτροπή Ήτρε και γνωρίζω ότι οι πανεπιστημιακοί φορείς συμμετέχουν και σε διεθνή και όχι μόνο ευρωπαϊκά δίκτυα. Ο άλλος λόγος είναι ότι τα πανεπιστήμια δεν είναι σημαντικά στα πλαίσια της ε, πρώτης και δεύτερης αποστολής τους ε, εκπαίδευση και έρευνα, αλλά και στην τρίτη αποστολή τους, δηλαδή την ανάπτυξη. Την ανάπτυξη ώστε να βελτιώνεται και να ολοκληρώνεται η επαγγελματική κατάρτιση της επιχειρηματικότητας συνολικά. Και σε αυτό θα πρέπει να συμμετάσχουν οι επιχειρήσεις ώστε να προχωρούμε στην ε, καινοτομία εκτός από τις θετικές επιστήμες και την εφαρμοσμένη τεχνολογία και στις κοινωνικές επιστήμες. Θα πρέπει λοιπόν να συζητήσουμε σχετικά με το πώς σήμερα τα πανεπιστήμια είναι εδαφικοί φορείς χωρίς να είναι δέσμοι του εδαφικού επίπεδου. Είναι πρωταγωνιστές, ηγούνται ε, αυτής της προσπάθειας στα πλαίσια αυτής της κρίσης που είναι και κρίση απασχόλησης που πλήττει τους νέους και επομένως αφορά άμεσα στα πανεπιστήμια που είναι και κρίση λοιπόν ε, ταυτότητας Χρειάζεται λοιπόν προσπάθεια όχι μόνο στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και της κατάρτισης. Ξέρετε ότι μας απασχολεί το θεματολόγιο το ευρωπαϊκό των νέων δεξιοτήτων και αυτό είναι ένα νέο πλαίσιο του οποίου πρέπει να εξετάσουμε, να αναρωτηθούμε τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερο, αλλά και τις λεγόμενες soft competence, τις άτυπες δεξιότητες, αυτές που αναπτύσσονται με την προσωπική εμπειρία. ώστε να έχουμε την εκκίνηση νέων επιχειρηματικών προσπαθειών με τη συνεργασία και την προσπάθεια των πανεπιστημίων. Ώστε να καλύψουμε αυτό το κενό που έχουμε σήμερα, το έλλειμμα που έχουμε των ε, δεξιοτήτων προκειμένου να μπορέσουν οι πανεπιστημιακοί φαρείς να δώσουν στην νεολαία τις δεξιότητες αυτές που είναι απαραίτητες για την κάλυψη θέσεων εργασίας και για την έρευνα. Είναι ευρύ το πεδίο. Ευχαριστώ όλους για τη συνεισφορά τους και θα πρότεινα και στην γραμματεία να συλλέξουμε όλες αυτές τις ε, συνεισφορές και να τις ε, δημοσιεύσουμε ε, γιατί πρόκειται για πολύτιμη δουλειά. Γνωρίζετε ότι οι χρόνοι που έχουμε για τις παρουσιάσεις είναι αρκετά περιορισμένοι και γι' αυτό το λέω. Θα δώσουμε λοιπόν σήμερα το λόγο στους ομιλητές μας και θα σας τους παρουσιάσω πρωτού ακούσουμε. Η κυρία Μάργκερ Μπρούς λοιπόν από το Πανεπιστήμιο του Ντάρμπι που θα μας μιλήσει για το σύγχρονο πανεπιστήμιο στον Ηνωμένο Βασίλειο και για την ενίσχυση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων τον ε, ρήτορα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης τον κύριο Μίτκα που είχα την τιμή να τον γνωρίσω. Του, του πρίτανε του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου λοιπόν, του κύριο Μίτκα, σχετικά με την ε, κρίση που αντιμετωπίζει η οικονομία και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας συναντηθήκαμε στην Ελλάδα σε μια δραματική στιγμή όπου εμείς ε, δώσαμε τη μάχη για να προστατεύσουμε την Ελλάδα να μην υπάρξει. Το Brexit, θυμάμαι και την έκκλησή του, την δραματική του έκκληση, ώστε να υπάρξει μια βοήθεια στο... και να διαδραματίσουμε κι εμείς ένα πιο σημαντικό ρόλο. Ο κύριος ε, Λόγγι, ε, πρίτανης ε, του Πολυτεχνείου των Μάρκε, τον κύριο Σεφτσικ, δεν ξέρω αν τον προφέρω σωστά, ε, καθηγητή του Πολυτεχνείου της Δρέσδης που θα μας μιλήσει για το ρόλο των πανεπιστημίων και των startup στην ε, ανάπτυξη περιφερειακών με στρατηγικών καινοτομία και τον κύριο Albert Πόιμερ που είναι project manager στο σύστημα CSB AG που θα μας μιλήσει για την ανώτη παιδεία στην περιφέρεια, στην Ήπεθρο συμβίωση μεταξύ Ακαδημίας και επιχειρήσεων. Ευχαριστώ λοιπόν εκ των προτέρων όλους τους συναδέλφους που είναι εδώ παρόντες. Θα έχουμε λοιπόν δύο τμήματα. Ένα πρώτο τμήμα παρουσιάσεων θα ανοίξει η κυρία Μπρούς και ο κύριος Μίτκας και μετά με ερωτήσεις και απαντήσεις από τα συναδέλφη, τους εκπροσώπους της Κομισιόν και ευχαριστούμε τους εκπροσώπους της εδώ και μετά θα έχουμε τους υπόλοιπους τρεις ε, παρουσιαστές ε, πάλι ε, μετά με ένα τμήμα Κυρία λοιπόν Μπρούς, σας δίνω το λόγο. Έχετε 10 λεπτά και με μεγάλο ενδιαφέρον περιμένουμε την παρουσίασή σας. Ευχαριστώ πολύ. Είναι μεγάλη μου χαρά που με προσκαλέσατε να παραβρεθώ και να συμμετάσχω σε αυτή τη δημόσια ακρόαση. Είναι πολύ καινοτόμο το να εξετάζουμε το ρόλο των πανεπιστημίων στην εξέλιξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Είναι μεγάλη μου χαρά λοιπόν που συναντώμε με, τον, ε, με την πρόεδρο ε, της Επιτροπής ε, Πολιτισμού και Ανάπτυξης, της κυρίας Κώστα, η οποία έχει ήδη δείξει πόσο πολύ την ενδιαφέρει και πόσο θέλει να συμμετάσχει σε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα που αφορά όλη την Ευρώπη. Το πανεπιστήμιο που εκπροσωπώ είναι ένα πανεπιστήμιο το οποίο έχει ως στόχο του την αριστεία, την ε, καινοτομία και βρίσκεται στην καρδιά του Ηνωμένου Βασιλείου σε μια περιοχή η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, είναι κέρια σημασίας ε, για την προηγμένη κατασκευή έχουμε ε, πάρα πολλές ε, μεγάλες ε, εταιρίες που βρίσκονται πολύ κοντά στο πανεπιστήμιο, ας πούμε την Toyota, την Rolls-Royce, την Bombardia. Οι αλυσίδες εφοδιασμού είναι εκεί. Σήμερα, σήμερα το πρωί μιλήσατε για τις δεξιότητες, την ανάγκη να, υπάρχει, να υπάρχουν οι ικανότητες. Αυτές που δίνουμε και εμείς στο Πανεπιστήμιο του Ντέρμπι, ώστε να έχουν οι φοιτητέ μας τις βέλτιστες ικανότητες ε, για να εξυπηρετήσουν ε, την ενδοχώρα, την περιοχή που εμείς εξυπηρετούμε. Εμείς ε, λοιπόν στέλνουμε από φύτους στην Rolls Royce για παράδειγμα. Βλέπουμε ότι η Rolls Royce έχει ανθρώπους από την περιοχή που απασχολεί και βλέπουμε το πανεπιστήμιό μας ως έναν καταλήτη της αλλαγής. Θέλουμε να εκπληρώνονται αυτές οι προηγμένες δεξιότητες. Θέλουμε να υπάρχει σωστή σύνδεση μεταξύ του ακαδημαϊκού χώρου και των επιχειρήσεων έτσι ώστε να προωθήσουμε την καινοτομία. Θα σας δείξω λοιπόν μια μελέτη περίπτωσης που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Πώς εμείς συνεργαζόμαστε και έχουμε κάνει με μια, μια εταιρική σχέση με άλλα πανεπιστήμια στην περιοχή. Προσπαθούμε αντί να ανταγωνιζόμαστε ο ένας τον άλλον να συνεργαζόμαστε, να δημιουργήσουμε ένα κεφάλαιο, μια αξία που θα χρησιμοποιηθεί στην περιοχή και να βρούμε τρόπους για να διευκολύνουμε τις εταιρείες να έρθουν σε επαφή μαζί μας και να συνεργαστούν, είτε πρόκειται για μικρές, ε, μικρομεσές ή μεγάλες επιχειρήσεις. Έχουμε λοιπόν αυτό το πανεπιστήμιο της επιχείρησης, όπως ονομάζουμε, το οποίο διασφαλίζει ότι οι φοιτητέ μας έχουν τα κατάλληλα προσόντα, τα εργαλεία για να εργαστούν στις επιχειρήσεις είτε της περιοχής μας είτε αλλού. Θα δείτε από τη διαφάνεια πόσο ισχυρή είναι αυτή η συνεργασία σε αυτή την περιοχή ε, του Ηνωμένου Βασιλείου. Έχουμε 146.800 φοιτητές και απασχολούμε πάνω από 17.000 άτομα ως όμιλος πανεπιστημίων δημιουργούμε 33.000 θέσει εργασία στην περιοχή των Midlands. Μέσα από την καινοτομία, ε, μέσα από τις επιχειρήσεις που συνεργαζόμαστε δημιουργούμε θέσεις εργασίας και έχουμε ένα ε, τζίρο 1,3 δις ε, λίρες το χρόνο. Ως ομάδα λοιπόν πανεπιστημίων έχουμε μεγάλη συνεισφορά. Η συνεργασία είναι θεμελιώδους σημασίας και την εκτιμούν οι επιχειρήσεις της περιοχής. Το Πανεπιστήμιο του Ντέρμπι έχει στο DNA του αυτά τα στοιχεία. Είναι η βασική μας αποστολή. Και υπάρχουν κάποιες αρχές που υποστηρίζουν αυτή την αποστολή. Είναι η οικονομική ανάπτυξη που υποστηρίζουμε για τις επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργαζόμαστε αλλά και για όλη την περιοχή. Συνεχώς έχουμε επαφή με τους ντόπιου ηγέτες, είτε απλούς πολίτες, είτε επιχειρηματίες, είτε ε, μέλη της κυβέρνησης και του ευρύτερου δημόσιου τομέα για να μπορέσουμε να επιτύχουμε τις προτεραιότητές μου ε, η Αντιπρίτανης επίσης ήταν στο, στο εξωτερικό και αυτό ακριβώς έδειχνε πόσο μεγάλη αξία έχει αυτή η συμμετοχή σε αυτό το πρόγραμμα για όλη την περιοχή, όχι μόνο για τον Τέρμπι. Δημιουργούμε λοιπόν ε, αποσχολησιμότητα, βελτιώνουμε την συγκράτηση των αποφύτων στην περιοχή Θέλουμε να έχουν πολύ καλές επιδόσεις και να διασφαλίσουμε ότι θα μείνουν στην περιοχή μας, θα φτιάξουν εκεί ε, μια σωστή σταδιοδρομία για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν το εργατικό δυναμικό της περιοχής, να φτιάξουν δικές τους επιχειρήσεις. Στο Πανεπιστήμιο θέλουμε να διασφαλίζουμε ότι έχουμε και τις βέλτιστες ακαδημαϊκές ικανότητες ε, που μας βοηθούν να συνεργαστούμε με τη Rolls Royce, την Bombardier, αυτές τις μεγάλες εταιρείες, να θέλουν δηλαδή να έχουν συνεργασία μαζί μας. Θέλουμε να προωθήσουμε την επιχειρηματικότητα γιατί θεωρούμε ότι αυτό για τους φοιτητές αυξάνει την απασχολησιμότητά τους. Ε, μπορεί να φτιάξουν οι ίδιοι εταιρείε ή να έχουν τα ταλέντα και τις δεξιότητες για να μπουν σε άλλες επιχειρήσεις και να φέρουν την αλλαγή εντός αυτού του ε, πλαισίου. Ως πανεπιστήμιο δηλαδή θέλουμε να δημιουργήσουμε πλούτο, εισόδημα. Ε, η αποστολή μας ε, και αυτό θα το συμμερίζονται και οι άλλοι φαντάζομαι του δικτύου μας είναι πολύ σημαντική και το θέμα είναι πώς την επιτυγχάνεις. Εμείς στο Πανεπιστήμιο του Ντέρμπι έχουμε αλλάξει και οι ίδιοι. Έχουμε μεταστρέψει την εικόνα μας έτσι ώστε να γίνουμε πιο ελκυστικοί για τις επιχειρήσεις, να θέλουν να συνεργαστούν μαζί μας και εμείς να μπορούμε να συνεργαστούμε μαζί τους. Συνεργαζόμαστε λοιπόν με τις εταιρείες για να δούμε εάν όντως ε, να διασφαλίσουμε ότι και το δικό τους προσωπικό είναι, έχει τις κατάλληλες δεξιότητες. κάνουμε μία εκπαίδευση ε, σε επιχειρηματικά ζητήματα. Επίσης έχουμε ε, τις εταιρείες που παίρνουν δικούς μας φοιτητές αλλά και ε, προγράμματα δικά μας για τους απασχολούμενους τους. Αυτοί λοιπόν που προέρχονται από μας χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας και μετά έχει να κάνει λοιπόν με μια εταιρική σχέση η οποία έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός εργατικού δυναμικού που έχει τη δυνατότητα να δημιουργηθεί να, δουλέψει σε αυτή τη βιομηχανία. Επίσης εξετάζουμε τις προτεραιότητες του τομέα, ας πούμε μεταφορά, χαμηλές εκπομπές αερίου, ε, αυξημένες ε, ε, απαιτήσει σε επίπεδο logistics. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι αυτά υπάρχουν. Θέλουμε να προβλέπουμε το μέλλον, να δούμε ποια θα είναι τα στοιχεία, οι δεξιότητες, ε, ακόμα και σε... Ε, όλο όχι μόνο σε επίπεδο γνώσης αλλά και σε επιθαρχικό επίπεδο για να μπορούν οι φοιτητέ να εξυπηρετούν τους σκοπούς, ε, να προσθέτουν αξία. Έχουμε επίσης ένα ταμείο επιχειρηματικών κεφαλαίων 17 εκατομμυρίων λιρών για να ενισχύσουμε την καινοτομία και θέλουμε να δημιουργήσουμε πάνω από χίλιες θέσεις εργασίας. Θέλουμε οι απόφοιτοί μας εκεί να απορροφηθούν. Δημιουργούμε μια διέξοδο για τις επενδύσεις μας, αν θέλετε. Μια διαρθρωτική χρηματοδότηση ε, μέσα από τα πλαίσια της, της κυβέρνησής μας και του περιφερειακού πακέτου ανάπτυξης. Ε, από το δικό μας λοιπόν πανεπιστήμιο έχουμε 10 εκατομμύρια επενδύσεων ε, που περνάνε σε επίπεδο χαμηλών εκπομπών και φτάνουν μέχρι τις μεταφοράς, τα logistics. Έχουμε 800 εταιρείες ε, που στην ουσία συνεργάζονται περίπου με, 400, με 4.000 άλλες μικρομεσαίες επιχειρήσεις για αυτό το στόχο. Ε, την καινοτομία δηλαδή και την ανάπτυξη των ε, δεξιοτήτων και τα κονδύλια που έχουμε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, αυτό το στόχο έχουν επίσης. Θέλουμε ε, οι απόφοιτοί μας να φτιάξουν startups ε, που μετά ε, θα στεγάσουν κέντρα καινοτομία και επιστήμης. Έχουμε πραγματικά επενδύσει σημαντικά στη δημιουργία υποδομής που θα βοηθήσει τις νεοσύστατες επιχειρήσεις να βρουν τα κονδύλια που θα τις βοηθήσουν να καινοτομήσουν. Επίσης δίνουμε και ε, υποστήριξη σε κλάστερς καινοτομίας. Για να δούμε τώρα πώς δημιουργούμε την αξία. Βλέπετε πώς η, η διαφάνεια αυτή δείχνει τον τρόπο που γεννάται η αξία και πώς αυτή προωθεί την καινοτομία. Και εδώ βλέπετε ένα διάγραμμα, αν θέλετε, της δομής που έχουμε στο Πανεπιστήμιο αυτή που, μας επιτρέπει να είμαστε ευέλικτοι. Έχουμε την μεταφορά γνώσης, συνεργαζόμαστε με εμείς ε, ως ε, ε, θεσμός πανεπιστημιακός με τις επιχειρήσεις. Θέλουμε αυτές οι επιχειρήσεις να έρθουν σε συνεργασία με το κέντρο, το Ινστιτούτο Καινοτομίας, για να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τις ε, δεξιότητες που προσφέρονται ε, για τις ανάγκες τους. Είναι μία προσέγγιση μεταφοράς γνώσης, αλλά είναι και πολύ ευέλικτη ταυτόχρονα. Εδώ ένα παράδειγμα πολύ καλό μεταφοράς γνώσης. Έχουμε την ε, πολύ προηγμένη τεχνολογία η οποία βοηθά τις επιχειρήσεις να καινοτομήσουν περαιτέρω. Ποιο είναι λοιπόν αυτό το επιχειρηματικό πανεπιστήμιο που θέλουμε να σας παρουσιάσουμε. Είναι ε, ένα πανεπιστήμιο που εξοπλίζει τους φοιτητές, τους, τους φοιτητές του να γίνουν και αυτοί καινοτόμοι. Οι επιχειρήσεις εντοπίζουν τα ταλέντα και έχουμε και ένα ταμείο επιχειρηματικών κεφαλαίων για τους φοιτητές ε, που επενδύει σε πολλά υποσχόμενες ε, αριστεύουσες επιχειρήσεις. Θέλουμε βέβαια αυτές οι εταιρείε να είναι ε, στην τοποθεσία αυτή, στην περιοχή μας δηλαδή, και να τις καθοδηγούν αυτά τα νέα ταλέντα. Για να συνοψίσω, εδώ θα δείτε κάποιους από τους βασικούς τρόπους που ξεκλειδώνουμε τη δυνατότητά μας να συνεργαστούμε με τις επιχειρήσεις. Είμαστε ευέλικτοι, επικεντρωμένοι, ο, επίσης ε, εξετάζουμε το μέλλον για να μπορούμε να προστατευτούμε από μελλοντικέ προκλήσεις. Προσπαθούμε να έχουμε ικανότητε υψηλή αξία. συνεργαζόμαστε μεταξύ μα έτσι ώστε οι άνθρωποι που βγαίνουν από εμά να μπορούν να εξυπηρετήσουν τους, σκοπούς που εμείς, σκοπούς εξυπηρετούμε. Επίσης υπάρχει μια αξία κεφαλαίου σημασίας που προωθεί την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. Στα κέντρα έρευνας ε, και τα Ινστιτούτα μας έχουμε εμπειρογνώμονες ειδικού ε, σε μια πλειάδα θεμάτων για να μπορούμε να επιλύουμε προβλήματα που περιβάλλουν τη μεταφορά γνώσης. Όμως, ε, γενικά να γνωρίζουμε την αποστολή του Πανεπιστημίου μας σε επίπεδο αξίας που είναι να κάνει τη διαφορά, να δώσει τα ταλέντα ε, τους ανθρώπους αυτούς που χρειάζονται οι επιχειρήσεις για να δημιουργήσουν από μόνες τους πλούτο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που σας ε, πίεσα ε, Ζητώ συγγνώμη που σας πίεσα λίγο για το χρόνο, αλλά πρέπει να σεβαστούμε τα χρονικά περιθώρια όλοι μας. Ευχαριστώ πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση και τώρα δίνω το λόγο στον πρίτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Περικλή Μίτκα, για το επόμενο θέμα, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μεταξύ των αποφύτων των πανεπιστημίων όταν η οικονομία βρίσκεται σε ε, δυσπραγία. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι εδώ, με εσάς κυρίες και κύριοι, και που απευθύνουμε στην Επιτροπή Πολιτισμού και Εκπαίδευσης. Αν διαβάσετε αυτό το τίτλο, ο στόχο είναι προφανής. Αλλά το πώς επιτυγχάνεται δεν είναι ίσως τόσο προφανές. 15 χρόνια ήμουν ε, μεταπτυχιακός και πανεπιστημιακός στις Ηνωμένες Πολιτείες και άρα ε, έχω την νοοτροπία του να είμαι σε επαφή με την οικονομία, με τις επιχειρήσεις σε διαρκή επικοινωνία μαζί τους. Ε, είμαι μηχανικός υπολογιστών. Όταν επανήλθα στην Ελλάδα το 2000 διαπίστωσα ότι στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στην Ελλάδα η κατάσταση είναι λίγο διαφορετική. Στην Ευρώπη δεν υπάρχει η ίδια αντιμετώπιση. Δεν ε, θεωρεί, δεν θεωρείται στην Ευρώπη ότι τα πανεπιστήμια πρέπει να είναι ατμομηχανές της ανάπτυξης. Διότι δεν είναι τόσο εύκολο να μεταφερθεί η τεχνολογία που παράγεται στα πανεπιστήμια στον ιδιωτικό τομέα. η κατάσταση ε, γίνεται ε, χειρότερη όταν κινείται κανείς από τον ε, βορρά προς τον νότο και από την δύση προς την ανατολή βέβαια με κάποιες εξαιρέσεις για τις οποίες το συγγνώμη. Πώς συνεργάζονται λοιπόν τα πανεπιστήμια και οι επιχειρήσεις όταν η χώρα είναι σε κρίση η Ελλάδα είναι σε κρίση εδώ και αρκετά χρόνια αν δείτε εδώ αυτή τη διαφάνεια, βλέπετε ότι μεταξύ του 2008 και του 2013 το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 25%. Περίπου όσοι ήταν η πτώση του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Μετά από 7 χρόνια λιτότητας έχουμε υψηλή ανεργία, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων σοβαρή αποεπένδυση, τρομερή μείωση των ξένων επενδύσεων, βαθιές περικοπές, ιδίως στην εκπαίδευση και ε, μαζική φυγή, διαρροή εγκεφάλων, που μπορεί να είναι βέβαια κέρδος για άλλες περιοχές της Ευρώπης και ευρύτερα. Έχουν αναφερθεί 200.000 απόφοιτοι ότι έχουν ε, φύγει από τη χώρα και είναι ε, ίσχυε πριν από 2.000 χρόνια. Σήμερα προσεγγίζουν τους 300, ε, τις 300.000. Παρ' όλα αυτά δεν υπάρχει έλλειψη ανθρωπίνου δυναμικού στην Ελλάδα. Μια έκθεση που έβγαλε το Σαντεφόπ την προηγούμενη εβδομάδα αναφέρει ότι υπάρχουν αναντιστοιχίες και λήψεις στην Ευρώπη των 28 μεταξύ δεξιοτήτων και αναγκών σε πέντε τομείς Σε ορισμένε χώρε βλέπουμε ότι υπάρχουν εξαιρέσει γιατί υπάρχει πλεόνασμα, πλεονάζονται δηλαδή με τα κατάλληλα προσόντα. Η Ελλάδα αναφέρεται σε τέσσερι από τι πέντε κατηγορίε. Οι Έλληνε νέοι έχουν γενικά μια ανοιχτή προσέγγιση. Θέλουν να βγουν από τη χώρα. 55% λένε ότι είναι διατεθειμένοι να φύγουν από τη χώρα και πολλοί φεύγουν. Είμαι πρίτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, Είναι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο τη χώρας. Αν δείτε που είναι η Θεσσαλονίκη, διαπιστώνετε ότι είναι πολύ κοντά σε πολλές ε, μεγάλες πόλεις των Βαλκανίων που επίσης προσπαθούν να αναπτυχθούν είναι μεγάλο πανεπιστήμιο, 78.000 φοιτητέ, πάνω από 78.000 φοιτητέ και το μεγαλύτερο ερευνητικό ίδρυμα τη ε, χώρας. Με πολλές ε, ερευνητικές δραστηριότητες, πάνω από 3.000 ε, νέοι εργάζονται σε ερευνητικά προγράμματα. Πέρα από τους τακτικούς ερευνητές εξαίρετη ποιότητα προπτυχιακών φοιτητών. Να σας δώσω παραδείγματα. Εδώ βλέπετε των διεθνών βραβείων που έλαβαν οι φοιτητές της Σχολής ε, Μηχανικών Υπολογιστών. Βλέπετε εδώ για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, Microsoft κτλ. Οι φοιτητέ μας λοιπόν ε, δουλεύουν πολύ και κάνουν και πολλές έξω πανεπιστημιακέ δραστηριότητες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη δημιουργία επιχειρήσεων αλλά δεν τα καταφέρνουν πολύ. Το αυτό ισχύει παντού στη Βόρεια Ελλάδα. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε λοιπόν ένα πολύ καλό κέντρο έρευνας και τεχνολογίας που αναφέρεται μεταξύ των ε, πρώτων 20 ιδρυμάτων αυτού του τύπου που λαμβάνουν δηλαδή τις περισσότερες επιδοτήσεις για έρευνα. Αλλά παρόλα αυτά δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε αρκετές θέσεις εργασίας για να κρατήσουμε αυτόν τον κόσμο. Όμως ε, ο λεγόμενος τριπλός έλικας, η συνεργασία μεταξύ των επιστημίων, ερευνητικών κέντρων, επιχειρήσεων του δυτικού τομέα και της κυβέρνησης, αρχίζει να, ε, να εξαπλώνεται. Έχει αλλάξει λοιπόν η νοοτροπία στην πόλη, που είναι μια πόλη ενός περίπου εκατομμυρίου κατοίκων, είναι και σημαντικό λιμάνι της Ελλάδας. Έχει τέσσερα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, όπου ε, φοιτούν γύρω στις 150.000 προπτυχιακοί και 30.000 μεταπτυχιακοί. Όλοι αυτοί λοιπόν συνεργάζονται και με το Δήμο, την πόλη, την περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας και τη ζώνη καινοτομία της Θεσσαλονίκη και άλλες ε, επιχειρήσεις, ε, την Τεχνόπολη, την ε, βιομηχανική ζώνη και άλλες επιχειρήσεις στην Βόρεια Ελλάδα. Μία πρόσφατη πρωτοβουλία είναι το λεγόμενο OK θες, είναι προθερμοκοιτίδα, όπου μικρές ομάδες φοιτητών, προσφάτων από τα κτλ. μπορούν να ανταλλάξουν ιδέες και να έρθουν σε επαφή με εγκαθιδρυμένες επιχειρήσεις. Κυρίως ασχολείται με ανάπτυξη λογισμικού. Επίσης υπάρχει η Τεχνόπολης, που είναι μια πρωτοβουλία των επιχειρήσεων ε, τεχνολογίας της πληροφορία στη Βόρεια Ελλάδα. Έχουν οργανώσει hackathon στα τελευταία χρόνια για να επιλέξουν τους καλύτερους αποφύτους και να τους προσλάβουν. Υπάρχει λοιπόν δραστηριότητα που έχει ως αποτέλεσμα σημαντικές εκδηλώσεις, Θεσσαλονίκη, χώροι κοινή εργασίας, δυνατότητες χρηματοδότησης από επιχειρήσεις κυρίως ε, του εξωτερικού. Έχουμε λοιπόν ορισμένα επιτεύγματα, εταιρείε λογισμικού για παράδειγμα που κάνουν έρευνα και ανάπτυξη μηχανολογικού εξοπλισμού που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και κάνουν τις πωλήσει και την εμπορία των προϊόντων, των προϊόντων τους στις ΗΠΑ. Αλλά ακόμη το χάσμα μεταξύ των δυνατοτήτων που υπάρχουν στην πόλη και των αναγκών του πληθυσμού, τόσο ώστε οι ιδέες τους για έρευνα να γίνουν προϊόντα, αυτό το χάσμα εξακολουθεί να υπάρχει. Το Πανεπιστήμιο έχει την υπηρεσία σταδιοδρομιών και απασχόλησης. Και έχει και μία μονάδα καινοτομία και επιχειρηματικότητα. Έχει και την υπηρεσία μεταφοράς τεχνολογία και δίνει συμβουλές σε νεοπαγεί επιχειρήσει, σε startup για πρώτη φορά. Θα κάνουμε μία έκθεση ερευνητικών δραστηριοτήτων στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε όλα τα πανεπιστήμια, πολυτεχνία και ερευνητικά κέντρα της χώρας για να παρουσιάσουν τα πρόσφατα αποτελέσματά τους στις ιδιωτικές επιχειρήσεις για ενδεχόμενη χρήση. Αυτό θα γίνει τον ερχόμενο Μάιο. Οι Πριτάνης και οι καθηγητές, ακόμη και οι πολιτικοί καταλαβαίνουν ότι τα πανεπιστήμια δεν θα έπρεπε απλώς να είναι νησιά απομονωμένα παροχής γνώσης ότι πρέπει να παίξουν ρόλο καταλήτη για την ανάπτυξη. Έχουμε λοιπόν υιοθετήσει αυτή την προσέγγιση, είμαστε σε επαφή με άλλες χώρες, είχαμε μια πρόσφατη ε, εκδήλωση που οργανώθηκε στην Βοστόνη όπου συμμετείχα μαζί με ηθήνοντες από την ζώνη καινοτομία της Θεσσαλονίκης προσπαθήσαμε να παρουσιάσουμε τη Θεσσαλονίκη και την Ελλάδα ως έναν κατάλληλο τόπο για ανάπτυξη λογισμικού. Θέλουμε λοιπόν να αξιοποιήσουμε και τις δυνατότητες της ελληνικής διασποράς. Υπάρχουν πολλές οργανώσεις, φορείς, ενώσεις ε, παντού στον κόσμο που προσπαθούν να μας βοηθήσουν, να βοηθήσουν την Ελλάδα να βγει από την κρίση. Έχουμε κάποια αποτελέσματα. Μας προτείνουν ορισμένοι, μας προτείνουν υποτροφίες, άλλοι συνεργασίες, εταιρικέ σχέσεις ή προσλήψεις. Και να καταλήξω με μια πρόταση που ίσως ε, θα άξιζε να την ε, προωθήσουμε. Οι καθηγητές στο Πανεπιστήμιο και οι ερευνητές παντού στον κόσμο διαφέρονται κυρίως και αξιολογούνται με βάση τις δημοσιεύσεις τους και την χρηματοδότηση για έρευνα. Τους ενδιαφέρουν λοιπόν οι αναφορές στις εργασίες τους στις, ε, σε, στα ερευνητικά περιοδικά. Δεν ενδιαφέρονται για το τι γίνεται η έρευνά τους από τη στιγμή που θα δημοσιευθεί. Ίσως θα μπορούσαμε να έχουμε ένα μεταβατικό δίκτυ επιχειρηματικότητας για να μετρήσουμε την ε, δραστηριότητα στον τομέα της επιχειρηματικότητας και την παραγωγικότητα, δηλαδή πατέντες, ε, παράγωγα προϊόντα, προϊόντα που πολλούνται, όλα λοιπόν αυτά που παράγονται στο πανεπιστήμιο και κατόπιν μπαίνουν στην αγορά. Γι' αυτό το λέω ε, μετάβασης, δίκτυ μετάβασης καλύτερα. Δεν προτείνω ότι οι πανεπιστημιακοί δεν θα πρέπει πλέον να αξιολογούνται με βάση πόσες εργασίες και πόσε αναφορές εργασίες εργασίε γίνονται. Αλλά Ίσως θα μπορούσε να υπάρχει και ένα βραβείο για υψηλό δίκτυ χρηματικότητας. Να υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Στην Ελλάδα ο ελέφαντας στο δωμάτιο είναι η πολιτική κρίση. Η πολιτικο-οικονομική κρίση. Αν δεν επανέλθει η χώρα σε μια ομαλή πορεία, δεν θα μπορέσουμε να προσελκύσουμε πολλές επενδύσεις. Αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Είναι μια πολύ σημαντική όχι μόνο παρουσίαση αλλά μαρτυρία σχετικά με την κατάσταση αυτή, το πλαίσιο αυτό είναι πολύ ενδιαφέρουσα η πρότασή σας και η δουλειά σας. Προτού δώσω το λόγο στους συναδέλφους, θα ήθελα να καλέσω τον εκπρόσωπο της ε, Κομισιόν, ε, τον κύριο Κρόουλη, επικεφαλής ε, της μονάδας της υπεύθυνη για θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Κώστα. Ζητώ συγγνώμη για αυτήν την έλλειψη κομψότητος. Θα ήθελα να έχω ακούσει τους άλλους ομιλητές πριν την παρουσίασή μου, αλλά πρέπει να αποχωρήσω γιατί έχω άλλες δεσμεύσεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εσάς κυρία Κώστα και τους συναδέλφους σας της Επιτροπής. Ε, συμμεριζόμαστε την εκτίμησή σας ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα, το ρόλο της επιχειρηματικότητας στην καινοτομία, την σχέση μεταξύ των πανεπιστημίων και των επιχειρήσεων των τοπικών και περιφερειακών δομών και φορέων. Είναι σημαντικά ζητήματα. Ε, θα ήθελα να κάνω αυτό που συχνά κάνουν οι εκπρόσωποι οι κομισιόν σε τέτοιες περιπτώσεις, να σας ενημερώσω σχετικά με κάποια, ε, κάποιες τρέχουσες διαδικασίες για να δούμε κατά πόσον συμπίπτουν με τα όσα ετώνησαν οι ε, ομιλητές, οι πρώτοι δύο και αυτοί που θα μιλήσουν και μετά. Από το 2008 ε, έχουμε ε, συστήσει ένα University Business Forum όπου είναι ένας χώρος συνύπαρξης συζήτησης των δύο αυτών πεδίων και εμείς προσπαθούμε να ε, ενεργοποιηθούμε ως διευκολυντές αυτής της συζήτησης. Να δούμε τι... ποια σημεία είναι κοινού ενδιαφέροντος. Αυτό γίνεται έχει γίνει πλέον μια παράδοση ολομελίας ε, τακτικά και μεταφερόμαστε εκτός από τις Βρυξέλλες σε διάφορα άλλα σημεία της Ευρώπης. Φέτος είχαμε τρία φόρουμ, ένα στη Βιέννη, ένα στη Φιλανδία και ένα στο Σαν Σεμπαστιάν, στην ε, χώρα των Βάσκων, στην Ισπανία. Ε, πρόκειται για ευκαιρίες όπου οι εκπρόσωποι των περιφερειών, των τοπικών αρχών, των πανεπιστημίων και των επιχειρήσεων συνομιλούν σχετικά με το τι συμβαίνει στο έδαφος της επιχειρήσης και τι άλλο χρειάζεται να συμβεί. Και νομίζω ότι έχει υπάρξει ένα πολύ ενδιαφέρον και παραγωγικό βήμα. Το περιέγραψα ως talking shop που είναι ίσως ένας ελαφρά ηρωνικός τρόπος, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουν προκύψει δύο συγκεκριμένες πρωτοβουλίες οι οποίες χρηματοδοτούνται από το Erasmus Plus, το οποίο γνωρίζετε. το σκεπτικό ήταν η ανάπτυξη ενός online μέσου που στην ουσία είναι ένα ερωτηματολόγιο, ένα εργαλείο αξιολόγησης ηλεκτρονικό όπου οι διάφοροι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αξιολογήσουν το βαθμό στον οποίο ο δικός τους φορέας είναι ανοιχτός στην επιχειρηματικότητα. Αυτό δημιουργήθηκε πριν από λίγα χρόνια και από τη δημιουργία του έχει αναπτυχθεί και χρησιμοποιείται πλέον από πάνω από 800 πανεπιστήμια, όχι μόνο στην Ευρώπη. Το ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι αυτή η αυτόνομη αξιολόγηση έχει οδηγήσει στην δημιουργία μιας κοινότητας. Μιας κοινότητας που ε, συζητά σχετικά με το τι χρειάζεται ώστε να υπάρχει πιο ενισχυμένη και πιο παραγωγική επιχειρηματικότητα και έτσι διευκολύνονται οι επαφές και οι συζητήσεις. Και μπορούμε να σας στείλουμε τα link γιατί έτσι μπορείτε να δείτε και να κατανοήσετε ποια είναι η διαδικασία και τι μπορεί να γίνει από μια μικρή επένδυση των 600.000 ευρώ που ήταν αυτή. Η δεύτερη συγκεκριμένη εξέλιξη που επίσης χρηματοδοτείται από το Erasmus Plus είναι μια δράση εταιρικών σχέσεων γνώσης που χρηματοδοτεί κονσόρτια επιχειρήσεων και πανεπιστημίων διασυνοριακά όπως πάντα συμβαίνει στο Erasmus ε, Plus για τη χρηματοδότηση νέου εκπαιδευτικού περιεχομένου για την παράδοση διδακτικών περιεχομένων με νέο τρόπο και με την παρουσία εκπροσώπων των επιχειρήσεων σε αυτές τις διαδικασίες τις μαθησιακές, τις εκπαιδευτικές. Ώστε να έχουμε, αν θέλετε, πρακτική εξάσκηση εντός του κόσμου των επιχειρήσεων. Έχουν χρηματοδοτηθεί περί τις 40 τέτοιες συγκεκριμένες δράσεις. Είναι πολύ νέο το μέσο και είναι δύσκολο να σας πω συγκεκριμένα τι έχει παραχθεί η ενδιάμεση αξιολόγηση θα μα πει περισσότερα σίγουρα, αλλά οπωσδήποτε έχει καταγραφεί η ενθουσιώδη συμμετοχή των ενδιαφερομένων και είναι άλλο ένα πλαίσιο που φέρνει πιο κοντά τα πανεπιστήμια και τις επιχειρήσεις. Συχνά όταν σκέπτονται οι αναλυτές την συνεργασία αυτή ε, θεωρούν ότι έχει να κάνει με την έρευνα δραστηριότητες στον πανεπιστημιακό χώρο, αλλά αυτό αφορά σε ένα ευρύτερο πεδίο για, την, για τον εμπλουτισμό του περιεχομένου που χρειάζονται οι ερευνητές και οι φοιτητέ. Κάτι ακόμα θα αναφέρω και γι' αυτό έλεγα ότι είναι κρίμα που μιλώ τώρα και όχι έχοντας ακούσει και την παρουσίαση του καθηγητή Σεφτσικ γιατί θα μιλήσει για το περιφερειακό επίπεδο της περιφερειακής στρατηγικής καινοτομίας αλλά αυτός ο συγκερασμός πανεπιστημίων και επιχειρηματικότητας στο φόρουμ οδηγεί πολύ γρήγορα, σχεδόν πάντα, στην ανάπτυξη περιφερειακών στρατηγικών. Όπως έγινε και στο Σαν Σεμπαστιάν. Ε, ιδιαίτερα στρατηγικές ευφυούς εξειδίκευσης, για παράδειγμα. Από την γάμα Delta Education and Culture ε, έχουμε συνεργαστεί με τους συνεδέλφους της γάμα Delta Regio ακριβώς σχετικά με αυτή τη στόχευση. Τι μπορούμε να συνεισφέρουμε και οι δύο στην ευφυή εξειδίκευση. Αλλά και πάλι εδώ μιλούμε για κάτι που βρίσκεται στα πρώιμα στάδια του, στάδια του αλλά οι συνάδελφοι από την Γενική Διεύθυνση Ρέγκιο μας λένε ότι βρίσκει κανείς περιφέρειες που προσπαθούν να οικοδομήσουν τέτοιες στρατηγικές χωρίς να συνομιλούν με τα πανεπιστήμια. Αυτό μας φαίνεται ε, ελληματικό, αν θέλετε, μη κατάλληλος τρόπος να προχωρήσει κανείς. Οπωσδήποτε αυτό είναι μια περιοχή στην οποία θέλουμε να δραστηριοποιηθούμε περισσότερο και τρόπος ναύρασης Μα έχει ζητήσει από τη Γενική Διεύθυνση να υποβάλουμε προτάσεις και ιδέες για το πώς μπορούμε να συνεισφέρουμε περισσότερο το 2017 ώστε να ενσωματώσουμε καλύτερα στα πλαίσια των στρατηγικών εφίους εξειδίκευσης τους πανεπιστημιακούς φορείς και ίσως την επόμενη φορά που θα έχετε εδώ τον Επίτροπο Πρόεδρε ε, να ήταν ενδιαφέρον θέμα να του υποβάλλετε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον εκπρόσωπο της Κομισιόν για αυτήν την ε, πολύ χρήσιμη συνεισφορά και να θυμίσω τα εξή. Εμείς ε, μάλλον μας έχει ήδη ανακοινώσει ο Επίτροπος ότι στις ερχόμενους μήνες θα έχουμε μια ανακοίνωση του εξυγχρονισμού του περιεχομένου της ε, ανώτατης εκπαίδευσης. Θεωρούμε λοιπόν ότι αυτή η ακρόαση θα είναι πάρα πολύ χρήσιμη και για όλους εσάς προκειμένου να καταλάβετε τι συζητείτε και τι ήδη συμβαίνει σε αυτό το επίπεδο. Και προκειμένου να ε, μπορέσουμε να εξετάσουμε και αυτό το θέμα, να το λάβουμε υπόψη. Το άλλο θέμα, που αργότερα το απόγευμα θα το συζητήσουμε και με τους συντονιστές, είναι μια πιο στενή συνεργασία με την Επιτροπή Ρέγγι, δηλαδή την Επιτροπή που ασχολείται με τις πολιτικές συνεχείς. Και θεωρώ ότι είναι πολύ σωστό αυτό που είπατε και πολύ χρήσιμο, έχοντας και την εμπειρία την περιφερειακή μου, μιλάω εδώ προσωπικά, είναι θέματα που συζητούσαμε με το δίκτυο το περιφερειακό. Δεν συμβαίνει πάντοτε αυτό, πράγματι, όπως σημειώσατε κι εσείς, και πρέπει να το σημειώνουμε αυτό στην εφαρμογή, στην υλοποίηση των προγραμμάτων και των προγραμμάτων συνοχής, μεταξύ άλλων. Λοιπόν, θα έδινε τώρα το λόγο στους ε, συναδέλφους που θέλουν να παρέμβουν. Λιμπάτσκα, Λιούαρ, Γραμματικάκης, Τρούπελ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους δύο για τις παρουσιάσεις σας. Συγγνώμη, έκανα λάθος και μίλησα πρώτος. Ναι, συγγνώμη. Οι κυρίες πρώτες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα σειρά παρουσιάσεων. Να αναφερθώ στα λόγια του Πρίτανη. Είπατε ότι το Πανεπιστήμιο θα πρέπει να είναι καταλήτης για την ανάπτυξη, την εξέλιξη. Ο καταλήτης όμως ε, απλώς επιταχύνει μια αντίδραση. Δεν αντικαθιστά τις, τα επιμέρους στοιχεία που λαμβάνουν μέρος σε αυτή την αντίδραση. Άρα, ε, γι' αυτό το λόγο έχουμε και ε, ανάγκη να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην ε, αλληλεξάρτηση των πανεπιστημίων και του οικονομικού περιβάλλοντος. Το πανεπιστήμιο, λοιπόν, πάντοτε βοηθάτε όταν έχει ένα ισχυρό οικονομικό περιβάλλον, όταν έχει ένα επικεντρωμένο κεφάλαιο. Όταν το κεφάλαιο είναι διασπαρμένο και βρίσκεται σε μικρές οντότητες και οι υπόλοιποι δεν ενδιαφέρονται για την καινοτομία, υπάρχει πρόβλημα. Άρα, πρώτο συμπέρασμα, η ανάπτυξη των πανεπιστημίων μέσω της καινοτομίας είναι ε, στην ουσία ε, μέρος ε, πολλών αλληλοσυμπληρωματικών δραστηριοτήτων, ξεκινώντας με το σχέδιο Juncker ή τον ορίζοντα 2020 που στην ουσία ε, βοηθούν και στην ενίσχυση λύσεων ακόμα και μέσα από φορολογικά κίνητρα. Τώρα για τον ορίζοντα 2020 που σύντομα θα αναθεωρηθεί να πω ότι επιτρέπει στα πανεπιστήμια να ενισχύσουν τις ερευνητικές τους δραστηριότητες και να τις αυξήσουν. Επίσης, ήμουν μέρος στο πρόγραμμα Marie Curie κοντόφσκα, το οποίο ενίσχυσε την ποιότητα των διδακτορικών στα πανεπιστήμια. Επιβεβαιώνεται αυτό που λέω. Και πώς εκποφελούνται τα ελληνικά πανεπιστήμια από τα, ε, τις επιχορηγήσεις μας στα πλαίσια του Οριζοντα 2020. Ευχαριστώ και τους δύο για τις παρουσιάσεις σας. Ε, να πω απλώς ότι είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένος που ε, το πανεπιστήμιο με το οποίο συνδέεται και το δικό μας γραφείο είναι εδώ. Φανταστείτε ποιο είναι. Ε, μιλήσατε για το συνεργατικό πανεπιστήμιο στο Τέρμπι. Τα πανεπιστήμια όμως μεταξύ τους ανταγωνίζονται και για τους καλύτερους φοιτητές πέρα από το να συναγωνίζονται και να συνεργάζονται. Πώς το συμβιβάζετε αυτό ε, για τη Θεσσαλονίκη, πώς αναπτύσσεται το αναλυτικό ε, πρόγραμμα, πώς έχει εξυγχρονιστεί πρόσφατα και πώς έχει ενισχυθεί αυτή η διαδικασία και επιταχυνθεί μετά την κρίση του 2008. Έχουν αλλάξει τα μαθήματα που παίρνουν οι Έλληνες φοιτητέ μετά την κρίση σε όλους τους επιστημονικούς τομείς. Και θα λέγατε επίσης ότι τα βασικά προσκόμματα στην επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα είναι διοικητικά ή είναι θέμα πολιτισμικό. Και αν είναι και τα δύο, να βασιστώ σε αυτό που είπε η Κομισιόν και να πω ότι η επιχειρηματικότητα δεν είναι απλώς η ίδρυση νέων σύστατων επιχειρήσεων. Θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας σχετικά με την ε, επιχειρηματικότητα ως ιδέα που ενισχύει ε, γενικά όλη τον ακαδημαϊκό χώρο, όχι μόνο τους συνήθεις ύποπτους, δηλαδή την ιατρική, την μηχανολογία κτλ. Τα λιγότερο συμβατικά θέματα της επιχειρημα... για την επιχειρηματικότητα, όπως είναι η ιστορία, η φιλοσοφία κτλ. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με την ενισχύση αυτή. Η κυρία Τρούπελ και μετά ο κύριος Ρωματικάκης, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ για τις παρουσιάσεις. Εγώ έχω μία ερώτηση για την κυρία Μπρούς. Όταν μας παρουσιάσατε την προσέγγισή σας και το τι προσπαθείτε να επιτύχετε μέσω αυτών των συστημάτων συνεργασίας, αναρωτήθηκα αν αντιμετωπίσατε κάποια προβλήματα και αν ναι, πώς τα υπερβήκατε και ποιος ήταν ο αντίκτυπός τους επί του μοντέλου, του προτύπου που αναπτύξατε. Παρακαλώ, κύριος Δηματικάκης. Ε, εγώ νομίζω κυρία Πρόεδρε ότι είναι πολύ σημαντική η σημερινή συνάντηση. Φαίνεται από τους ομιλητές, ε, φαίνεται από το ικανοποιημένο σας χαμόγελο, αλλά κυρίως φαίνεται από το ότι νομίζω ότι πριν από 20 χρόνια οι φοιτητέ στην Ελλάδα και παντού σε όλες τις χώρες της Ευρώπης είχαν ένα εύκολο δρόμο σπούδαζαν, έβρισκαν εύκολα δουλειά. Ήταν ένα ιδανικό που εύκολα ικανοποιούσαν οι χώρες. Σήμερα τα ποσοστά ενεργείας των νέων τα έχω σημειώσει γιατί όσο και να τα διαβάζω δεν τα πιστεύω. Στην Ελλάδα βέβαια που έχει τη θλιβερή πρωτιά είναι 42,7%. Στην Ισπανία δεν πάει πίσω 42,6%. Ιταλία 37% και συνολικά στην Ευρωζώνη 20,3 συνολικά με τις πλούσιες χώρες μέσα. Είναι απίστευτο. Και παρόλα αυτά η Ευρώπη κινείται πάρα πολύ αργά στο να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα, εάν αντιμετωπίζεται. Εγώ επειδή δεν προσπαθώ να μην καταχραστώ ποτέ το χρόνο, που είναι πάντα λίγος και για τους ομιλητές, θα κάνω μόνο μία παρατήρηση και δύο πολύ απλές ε, επισημάνσεις. Προς την κυρία Μπρούς πρώτα-πρώτα. Με εντυπωσίασαν όσα είπε για το Πανεπιστήμιο που δεν το ξέρω από κοντά, παρόλο που δέκα χρόνια της ταπεινή ζωής μου τα πέρασα στην Αγγλία. Δηλαδή νομίζω ότι μας δώσατε μια πολύ ιδεώδη εικόνα, μακάρι να είναι έτσι. Εφτά πανεπιστήμια συνεργάζονται, είπατε. Σε ποια βάση συνεργάζονται. Εγώ δυσκολία έχω να δω δύο-τρία πανεπιστήμια να συνεργάζονται και κυρίως αυτό που με φόβησε και μπορεί να κάνω λάθος είναι ότι από όσα είπατε φαίνεται να παραμερίζεται τελείως αυτό το ακαδημαϊκό πνεύμα που είναι η ανάσα των πανεπιστημίων, η αγάπη των πανεπιστημίων, ο τρόπος ζωής τους προς όφελος κάποιων ας πούμε τι θα μπορούσε να διδάξει ένα πανεπιστήμιο όπως είπατε για να συνεργαστεί με τη Rolls Royce. Φαντάζομαι λοιπόν το επίτευγμά σας είναι πολύ σπουδαίο. Δεν θέλω να το αναιρέσω αλλά θα ήθελα να μου πείτε λίγα πράγματα παραπάνω. Και μου φαίνεται και πρωτοποριακό στο βαθμό που αυτή η συνεργασία επιτυχάνεται όπως μας περιγράψατε. Βέβαια ο κύριος Πρίτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ε, πρέπει να υπερηφανεύεται γιατί σε μια χώρα που βρίσκεται υποκρίση ε, καταφέρνει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το ξέρω από κοντά, το ξέρει όμως και η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Ε, εγώ είχα την κακή τύχη να είμαι έξι χρόνια στη θέση του στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης ως Πρίτανης, αλλά υπό πολύ καλύτερες συνθήκες. Και θα ήθελα να το ρωτήσω αυτό το αιώνιο ερώτημα. Η σχέση των πανεπιστημίων στην Ελλάδα με την πολιτική εξουσία δεν ήταν ποτέ καλές. Τουλάχιστον στη δική μου εποχή. Ελπίζω σήμερα να είναι καλύτερες. Η πολιτική εξουσία δηλαδή στην Ελλάδα αλλά και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, τα ακούμε σήμερα, με έμεσο ή άμεσο τρόπο προσπαθούν να επέμβουν στην αυτοτέλεια των πανεπιστημίων, άρα στον κύριο σκοπό της ε, υπάρξεώς του. Και δεύτερο θα ήθελα να ρωτήσω το φίλο κύριο Πρίτανη και όσοι τολμούν να δώσουν μια απάντηση, τέλος πάντων ε, τι περιμένουν τα πανεπιστήμια της Ευρώπης, των οποίων οι εκπρόσωποι είναι εδώ σήμερα, από αυτή την Ευρώπη που όλο λέει ότι πρέπει να αλλάξει αλλά δεν μου φαίνεται ότι αλλάζει και πάρα πολύ. Αυτά κύριε Πρίτανη και κυρία Πρόεδρε. Είναι μια περίπλοκη ερώτηση προκειμένου να απαντηθεί σε λίγα λεπτά. Εν πάση ελπίζω ότι χάρη στην προετοιμασία μας ε, θα μπορέσετε, θα είστε σε θέση να απαντήσετε λέει η Πρόεδρος. Κοιτάξτε. Ο ε, ορίζοντας 2020 είναι πολύτιμος, απαραίτητος. Ε, χρηματοδοτεί και επιτρέπει τη συνεργασία και τη διερεύνηση νέων δυνατοτήτων για συγκεκριμένα έργα. Ε, είναι λοιπόν ουσιώδες. Το Μαρί Curie κατά την άποψή μου και είχαμε εμπειρία, με αυτό έχει βελτιώσει την ποιότητα των διδακτορικών ερευνών ε, και έχει επιτρέψει σε περισσότερους να συμμετάσχουν σε αυτό το επίπεδο των σπουδών και είναι και αυτό πολύ καλό. Για τις νεοσύστατες ε, επιχειρήσεις, τα startups, για μένα το θέμα αυτό είναι σχεδόν αποτέλεσμα του να έχει κανείς ένα ε, πνεύμα επιχειρηματικότητας που είναι βαθιά ριζωμένο στην πανεπιστημιακή παιδεία. Στη δική μας περίπτωση είναι περίπου στο DNA μας να είμαστε καινοτόμοι και ε, ως προς την επιχειρηματικότητα για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, ε, για την έρευνα, ε, για νέες εισαγωγές και θεραπείες. Ανοίγει παντού δυνατότητες για τους αποφύτους να δραστηριοποιούνται σε νέα παιδεία, το οποίο είναι εξαιρετικό. Για την ε, Midlands, αυτό είναι κάτι καινούριο. Ε, έχουμε πολλές συζητήσεις σχετικά με τις αμοιβέ ανάγκες και το οποίο ασχολείται και με κάποιες, ε, αν θέλετε, τον ανταγωνισμό, τον επιθετικό ανταγωνισμό που ενδεχομένως υφίσταται σε κάποιες περιοχές. Ακόμα προσπαθούμε να αναπτύξουμε το modus operandi και κάποιε θεματικέ πιο συγκεκριμένε επί των οποίων ίσως να χρειάζεται να έχουμε καλύτερη πρόσβαση σε δυναμικό ή σε υποδομές στο σύνολο των πανεπιστημίων παρά μεμονωμένα. Και επιτρέπει και αναγνώριση των, του συνόλου, αν θέλετε, των πανεπιστημίων μέσω μια διαδικασία που είναι σχεδόν σαν αναγνώριση σήματος, brand name. Yes, I would like to ask uh, because my question is not answered. Ναι, δεν απαντήθηκε όμω η ερώτησή μου. Υπήρξαν προβλήματα. Θα ήθελα να μάθω τι προβλήματα υπήρξαν. Ε, ναι, μα είναι νέες αυτές οι τερικές σχέσεις. Και άρα είμαστε ακόμη σε περίοδο χάριτος. Αλλά δεν είναι απλώς πανεπιστημιακή φορείς, είναι και τοπικές αρχές, οι θύνοντες της τοπικής κοινωνίας, εξετάζουμε τις προτεραιότητες μας για ολόκληρη την περιοχή. Δεν είναι μόνο πανεπιστημιακοί, είναι και άλλοι. Συμμετέχουν επιχειρήσεις παντού από όλη την περιοχή. Για παράδειγμα, μπορούμε να ασχοληθούμε με την αλυσίδα εφοδιασμού. Έχουμε μια ομάδα, τη οποία ηγείται η Rolls Royce, άρα είναι μεικτή ομάδα για να εξετάσει τις περιφερειακές ανάγκες πέρα από τις ανάγκες των πανεπιστημίων. Και ίσως να βοηθάει αυτό λόγω της φύσης εταιρικής σχέσης ούτω ώστε να εστιάσουμε ευρύτερα. Επηρεάζει ε, το πρόγραμμα σπουδών επειδή τέθηκε το ερώτημα γιατί φυσικά θέλουμε στόχος μας να είναι να, να εμπλουτίσουμε τα πανεπιστήμια μας, να εμπλουτίσουμε το περιεχόμενο των σπουδών μας, την έρευνά μας, ε, τη διδασκαλία μας, ακριβώς ε, έχοντας επαφή με την ευρύτερη κοινωνία. Ευχαριστώ πολύ. Ξεκινώντας με το πώς υποφελούνται τα πανεπιστήμια από την έρευνα. Στην Ελλάδα τα πανεπιστήμια είναι δημόσια, οπότε δεν έχουν δίδακτρα. Παίρνουν χρήματα από το κράτος και από ερευνητικά προγράμματα. Θα σας δώσω κάποια νούμερα. Το 2009 το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο έλαβε περίπου 44 εκατομμύρια λειτουργικά ε, ε, για τα λειτουργικά έξοδα από την κυβέρνηση και περίπου 35 εκατομμύρια για έρευνα. Το 2015-16 έλαβε 12 εκατομμύρια από την κυβέρνηση για μεγαλύτερο αριθμό φοιτητών και δημιούργησε 50 εκατομμύρια σε έρευνα. Τα ερευνητικά προγράμματα είναι στην ουσία η ζωοδόχος πηγή για τα πανεπιστήμια που δεν έχουν αρκετή υποστήριξη από το κράτος βέβαια. Ο τρόπος που είναι διαρθρωμένα στην Ευρώπη στην ουσία απαιτεί τη συνέργεια μεταξύ πανεπιστημίων και εταιριών. Τα κέντρα ερευνών είναι πάρα πολύ καλά για τη δημιουργία αυτής της επιχειρηματικής ε, νοοτροπίας, όμως παρόλα αυτά δεν είμαστε πολύ επιτυχημένοι γιατί όταν τελειώνει το project τα αποτελέσματά του ξεχνιόνται. Ε, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παράγει δηλαδή. Θα μπορούσαμε να τα πάμε καλύτερα. Πώς έχει αλλάξει το αναλυτικό πρόγραμμα στην Ελλάδα πολύ λίγο. Και θα σας πω γιατί. Γιατί τα τελευταία 7-8 χρόνια υπήρξε ε, στην ουσία μεγάλο πρόβλημα στα διάφορα τμήματα επειδή χάνουμε καθηγητές είτε γιατί βγαίνουν στη σύνταξη και δεν αντικαθίσταται είτε γιατί φεύγουν. Ε, για τους επιστημονικούς λοιπόν τομείς αυτούς ε, είναι πολύ δύσκολο να αλλάξεις το αναλυτικό πρόγραμμα όταν δεν έχεις νέους ανθρώπους να τροφοδοτούν τις εργασίες του Πανεπιστημίου. Επίσης, οι επιλογές ε, των φοιτητών άλλαξαν. Πέρασαν από δουλειές που οδηγούν σε κυβερνητικές θέσεις, σε θέσεις μάλλον στο δημόσιο, σε άλλες ε, επιδιώξεις, να δουλέψουν δηλαδή στη βιομηχανία. Είδαμε δηλαδή αλλαγή στις επιλογές τους. Τώρα, ποιοι είναι οι αγοραστές τα προσκόμματα στις συνέργειες μεταξύ των ε, επιχειρήσεων και των πανεπιστημίων. Ανάλογα με το νομικό σύστημα της άλλης χώρας υπάρχει αυτό το πρόβλημα, όπως είπε και ο κ. Γραμματικάκης, και βέβαια είναι και θέμα γραφειοκρατίας και νοοτροπίας. Στην Ελλάδα για χρόνια είχαμε μια νοοτροπία που έλεγε ότι τα πανεπιστήμια είναι τελείως διαφορετικά από την ε, βιομηχανία, από τις επιχειρήσεις και δεν πρέπει μεταξύ τους να συνδιαλέγονται. Αυτή η νοοτροπία έχει αλλάξει και είμαι σίγουρος ότι ε, αλλάζει πολύ πιο γρήγορα στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες πηγαίνοντας από το βορρά στο νότο και από την ε, δύση προς την Ανατολή. Εμείς ε, φυσικά δεν είμαστε ούτε στη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών, ούτε στη θέση του Ισραήλ. θα μπορούσαμε να πάρουμε κάποια μαθήματα από αυτούς, ειδικά η Ελλάδα και χώρες σαν και αυτή. Για τον κύριο Γραμματικάκη, κύριε καθηγητά, συμφωνώ μαζί σας πλήρως. Ε, ε, μας πνίγει η κυβέρνηση στα πανεπιστήμια εδώ και χρόνια, ε, γιατί προσπαθούν να ελέγξουν κάθε μικρή πτυχή της λειτουργίας μας. Είναι δύσκολο. Και αυτό έχει επιδεινωθεί από το γεγονός ότι αλλάζει η νομοθεσία σχεδόν σε μηνιαία βάση τα τελευταία δύο χρόνια. Είναι δύσκολο λοιπόν ε, να βασιστούμε σε αυτήν. Ε, τι περιμένουν τώρα τα πανεπιστήμια από την Ευρώπη. Τι να πω πάντοτε θεωρούσα ότι τα πανεπιστήμια θα έπρεπε αυτά να υποδείξουν στην Ευρώπη προς τα που να κατευθυνθεί. Αυτοί έχουν τον κόσμο, την εμπειρογνωμοσύνη, τουλάχιστον αυτά θα έπρεπε να την αναπτύσσουν. Εγώ, όπως σας είπα, είμαι... Ε, ε, μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών. Αυτά τα πανεπιστήμια που δεν δημιουργούν καινούργια γνώση θα φανιστούν. γιατί οι φοιτητές μπορούν, μπορούν πλέον να μαθαίνουν με πολλούς τρόπους, όπου θέλουν, όποτε θέλουν. Δεν χρειάζονται μια τυπική εκπαίδευση μέσω πανεπιστημίου. Ένα πανεπιστήμιο που δημιουργεί νέα γνώση όμως θα παραμείνει ως βασικό ίδρυμα γνώσης. Τα πανεπιστήμια λοιπόν παραμένουν χρήσιμα, χρειάζονται την υποστήριξη της Ευρώπης, ακόμα και οι ανθρωπιστικές επιστήμες, όπως ανέφερε κάποιος, αλλά θα αλλάξουν τα πανεπιστήμια. Θα πρέπει να αλλάξουν. Αυτό το συμπέρασμα είναι πολύ όμορφο, νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι και είναι πολύ σημαντική ευθύνη και για τα πανεπιστήμια αλλά και για τις κυβερνήσεις και για τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε όλα αυτά να μπορέσουν να γίνουν με τη μέγιστη και η υπευθυνότητα και η ελευθερία ώστε να επιτύχουμε επιτέλους μια ανάπτυξη που να είναι βιώσιμη και που να συνδέεται με την καινοτομία, τη γνώση ε, και να συνοδεύεται και από την απαραίτητη κοινωνική προστασία. Σας ευχαριστώ λοιπόν και θα ζητούσα από τους επόμενους τρεις καθηγητές, το επόμενο πάνελ, να ζητήσω συγγνώμη από τον συνάδελφο Λίουερ ελπίζω να μας επιτρέψει αυτό το πλαίσιο του Brexit ε, να συνεχίσουμε τη συνεργασία ε, και να υπάρξει μια θετική κατεύθυνση για τις, για τις αποφάσεις που θα ληφθούν στη χώρα σας σχετικά με την ερευνητική δραστηριότητα των πανεπιστημίων. Σας ευχαριστώ και υποδέχομαι τους τρεις επόμενους καθηγητές Λοιπόν, αυτό είναι το επόμενο πάνελ των ομιλητών μας. Ο κύριος Λόγκη, εις όπως είπα ήδη, του ε, Πολυτεχνείου των Μάρκε από την Ιταλία, από την Αγκώνα. Και είμαι βέβαιο ότι εκφράζω όλους τους συναδέλφους ε, όταν δίνω ε, ευχές και εκφράζω πραγματικά την συμπάθεια όλων και τη συμπόνια όλων σχετικά με τα θύματα και τις ζημιές ε, του σεισμού στην ευρύτερη περιοχή. Παρακαλώ κύριε Λόγγι για την παρουσίασή σας. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Το δικό μας πανεπιστήμιο ε, βρίσκεται στις ε, Μάρκε, που είναι η 8η παραγωγός περιφέρεια της Ευρώπης. Πολύ μικρή περιφέρεια, αλλά ακόμα σε θέση να παράγει σε επίπεδα ποσοτικά πολύ σημαντικά. Άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι παρά του 1.800.000 κατοίκους έχουμε 552.000 επιχειρήσεις. Δηλαδή έχουμε μια διάχυση της επιχειρηματικότητας αν θέλετε πολύ μεγάλη και κατά μέσον όρο για κάθε χίλιους κατοίκους έχουμε 100 και άνω επιχειρήσεις. Επομένως, αν θέλετε, υπάρχει μια δραστηριότητα επιχειρηματική που ιστορικά έχει αναγνωριστεί εδώ και πολλά χρόνια. Και έχουμε να κάνουμε με επιχειρήσεις που ξεκινάνε από ένα πολύ απλό επίπεδο. Αυτό που εμείς προσπαθούμε να κάνουμε ως πανεπιστήμιο είναι να δώσουμε κίνητρα επιχειρηματικότητας στις περιφέρειες, να πλησιάσουμε το πεδίο αυτό προς τη γνώση και να διευκολύνουμε τους καινούριου τρόπους δημιουργίας σύστασης επιχειρήσεων, όχι μόνο ως προς τις οικονομικές και εμπορικές στοιχές τους, αλλά σε επίπεδο γνώσης, ώστε να μπορούν αυτές οι επιχειρήσεις να είναι βιώσιμες, να αναπτύσσονται, να αξιοποιούν νέα στοιχεία. Αυτός είναι ο ρόλος που πρέπει να αναλαμβάνει ένα πανεπιστήμιο. Εγώ πιστεύω ότι η Ευρώπη χρειάζεται έντονα την επιχειρηματικότητα, χρειάζεται τις καινούργιες γενιές πρέπει να ενισχύσουμε το πλαίσιο και τη δυνατότητα αυτή, την δημιουργικότητα που μπορεί να οδηγήσει σε νέες ευκαιρίες, σε νέες επιχειρήσεις. Βρισκόμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο ε, και πρέπει να βοηθήσουμε τους νέους να εφεύρουν θέσεις απασχόλησης για τους ίδιους και για τους υπόλοιπους. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και στο έδαφος, γιατί είμαστε ένα πανεπιστήμιο, ένα πολυτεχνείο που είναι βαθιά ριζωμένο στον τόπο του και προσπαθούμε να εμπνεόμαστε από τις ιδιαιτερότητες ε, τις εδαφικές τις δικές μας. Προσπαθούμε λοιπόν ε, να έχουμε παραδοτέα σε επίπεδο γνώσης, γιατί θεωρούμε ότι η προσθέμενη αξία στις επιχειρήσεις σήμερα είναι εκείνη που βασίζεται ακριβώς στη γνώση, στην έρευνα, στις εξειδικευμένε γνώσεις που σωρεύονται εντό του Πανεπιστημίου. Όπως ελέγχθηκε στο προηγούμενο πάνελ. Αυτό πρέπει να αξιοποιήσουμε. Και πώς μπορούμε να το κάνουμε. Εδώ ήδη αναφέρθηκαν διάφορα πρότυπα, διάφορα κέντρα ερεύνης που συνεργάζονται μεταξύ τους. Αναφερθήκαμε σε μια δικτύωση ή καθοδήγηση της επιχειρηματικής προσπάθειας των νέων. Συχνά αυτό γίνεται μέσω της αξιοποίησης της έρευνας ώστε να πάμε στη δημιουργία startup, νεοσύστατων επιχειρήσεων με απλά βήματα. Και αυτό είναι το πρώτο σκαλοπάτι προς την κατεύθυνση αυτή, αλλά δεν φτάνει. Πρέπει μετά να απτύξουμε όλες εκείνες τις ε, διασυνδέσεις, τους συσχετισμούς που είναι απαραίτητες προκειμένου να προχωρήσει αυτή η καινούργια ιδέα. Ε, στην προηγούμενη προσχέση ακούσαμε την σημαντική παρουσία του, του venture capitalism, ε, την πολύ σημαντική στην δημιουργία των νέων επιχειρήσεων. Επομένως, πέραν της αξιοποίησης της έρευνας αυτής και της ε, ανταλλαγής μεταξύ των δύο κόσμων, χρειάζεται και αυτός ο σχετισμός. Ποια είναι λοιπόν η στρατηγική που χρησιμοποιήσαμε εμείς ώστε να βοηθήσουμε αυτές τις δράσεις. Το πρώτο είναι αυτό που εμείς αποκαλούμε ανταλλαγή εμπειρίας. Την επιμόλυνση της εμπειρίας όπως την αποκαλούμε. Προσπαθούμε να πάμε σε δράσεις καινοτόμες. Υπάρχει καινοτομία στην καθημερινή ζωή μας. Μπορούμε να κάνουμε πάντοτε καλύτερα αυτό που κάναμε από χτες. Αλλά το μέλλον που αναζητούμε δεν είναι αυτό απλώς χρειάζεται σημαντική καινοτομία, ριζοσπαστική καινοτομία και επομένως χρειάζεται εμπειρι... Ε, ε, ε, σύγκριση των εμπειριών μεταξύ των διάφορων φορέων. Σύγκριση της όρευσης των εμπειριών. Έχουμε λοιπόν δημιουργήσει ένα εργαστήριο ένα εργαστήριο στο οποίο οι, διάφορες, οι διαφορετικές μάλλον ιδέες συγκρίνονται και αλληλοενισχύονται. Αυτό λοιπόν το έχουμε ονομάσει Contamination Lab, που είναι ένα εργαστήριο στο οποίο η κεντρική ιδέα, ο κεντρικός άξονας είναι ακριβώς αυτή η αλληλοεπιμόλυνση με τις ιδέες των διαφορετικών φορέων, των φοιτητών, των διαφορών τμήματων, σχολών και όλα αυτά σε διάφορα επίπεδα. Πρώτο, δεύτερο και τρίτο επίπεδο ε, μάθησης και προσπαθούμε να έχουμε και διασυνδέσεις με τον κόσμο των επιχειρήσεων ώστε κάθε περιφέρεια να δημιουργεί τη δική της ευφυή εξειδίκευση έτσι έχει κάνει και η περιφέρεια ε, των Μάρκε ώστε να μπορούμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί ακριβώς στην εξειδικευμένη αυτή κατεύθυνση που έχουμε επιλέξει. Και από εκεί και πέρα χαράζουμε την πορεία που χρειάζεται προκειμένου να συλλέξει κανείς την απαραίτητη εμπειρία, τις απαραίτητες δεξιότητες για την επίλυση των προβλημάτων, για ε, μια πραγματική ικανότητα επιχειρηματικότητας, αλλά και την ε, επικοινωνιακή ικανότητα που είναι θεμελιώδες στοιχείο της επιτυχίας στις επιχειρήσεις. Ε, χρειάζεται να επικοινωνούμε σωστά, δηλαδή να διαχέουμε αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε με αποτελεσματικό, με θετικό τρόπο. Έχουμε δημιουργήσει χώρους λοιπόν μαζί με το εργοστήριο αυτό, κλασικές αίθουσες αν θέλετε εκμάθησης και το διατηρούμε ανοιχτό ή δυνατόν σε κάθε ώρα της ημέρας, γιατί πρέπει να είναι ο, δημιουργικός, ο δημιουργικός αν θέλετε, κοινό τόπος. Ε, και το πιο σημαντικό, εμείς επιχειρήσαμε αυτό να το ξεκινήσουμε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Ουρμπίνο και της ε, Ματσεράτα, που είναι πανεπιστήμια ουμανιστικών σπουδών, ε, το δικό μας είναι πολυτεχνείο, προσπαθούμε λοιπόν να αναμίξουμε να αναμίξουμε τα διάφορα προγράμματα για να βλέπουμε, για να έχουμε μια προσέγγιση συνολικότερη. Εμείς ε, περιμένουμε να αναπτύξουμε μηχανικούς τις νέες τεχνολογίες. Θα περίμενε κανείς δηλαδή την ανάπτυξη των ρομπότ, αλλά βλέπουμε ότι οι σημαντικότερε καινοτομίες προέρχονται από τον κόσμο της ιατρικής και της γεωργίας. τη εξειδικευμένη γεωργίας. Από εκεί και πέρα βεβαίω και έχουμε ηλεκτρονικούς μηχανικούς, ε, οικονομολόγους. Όλοι αυτοί συνεισφέρουν ε, και ενισχύουν την ιδέα. Αλλά οι πιο σημαντικές ιδέες έχουν προέλθει από σπουδαστέ, που δραστηριοποιούνται σε τομεί πολύ διαφορετικού από εκείνου. που συνήθως αποκαλούμε ευφύ εξειδικεύση. Επομένως, αυτό που δημιουργήσαμε τελικώς με το εργαστήριο αυτό είναι η κατάργηση, αν θέλετε, σε κάποιο επίπεδο, των διαχωρισμών των προγραμμάτων μεταξύ τμήματων, μεταξύ σχολών, μεταξύ οικονομολόγων, φιλοσόφων, μηχανικών κτλ. ώστε να κινηθούμε, να καταφέρουμε αυτά τα αποτελέσματα που εμείς τα θεωρούμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Επιχειρήσαμε δηλαδή να εξωθήσουμε βία σχεδόν τη διαφορετικότητα. Γιατί μόνο από τη διαφορετικότητα ε, μπορούν να προκύψουν απρόβλεπτα, απρόβλεπτες νέες ιδέες, απρόβλεπτη καινοτομία. Κάτι δηλαδή που την προηγούμενη μέρα κανείς δεν περίμενε ότι θα συμβεί. Και αυτό είναι που χρειαζόμαστε για να ενισχυθεί όλο το πλέγμα της επιχειρηματικότητας. Ε, όπως σας έλεγα έχουμε μία επιχείρηση ανά 10 κατοίκους. Πρέπει να μεταφέρουμε λοιπόν γνώση και αυτό πρέπει να κάνει το Πανεπιστήμιο προς τον κόσμο των επιχειρήσεων. Άρα λοιπόν συνοψίζοντας θα έλεγα ότι το C-Lab μας, το Contamination Lab όπως έλεγα, είναι ένα ευρωπαϊκό πρότυπο συνδιαλλαγή συζήτησης συν, ομαδικής θα έλεγα ερευνητικής δραστηριότητας που αναζητούμε την καινοτομία από τη διαφορετικότητα όπως σας έλεγα, από την ποικιλία, από την σύγκριση μεταξύ διαφορετικών σχολών, τομέων, ειδικεύσεων. Γιατί θεωρούμε ότι αυτός είναι ο δρόμος που θα επιτρέψει στην Ευρώπη να συνεχίσει να αναπτύσσεται και να διαχέει το, δικό, το της πλούτο και τα δικά της μηνύματα. Εγώ, αν θέλετε, και προσωπικά ε, το υπερασπίζομαι αυτό σαν κεντρική ιδέα, αλλά θα έλεγα και όλοι οι σπουδαστέ μας, διότι η Ευρώπη είναι φτιαγμένη από πολλές διαφορετικότητες. Και πρέπει να τις αξιοποιήσει αυτές τις διαφορετικότητες, ώστε να συνθέσει μέσω αυτών δυνατότητα γιατί είναι οπωσδήποτε ένα πλεονέκτημα που έχουμε. Και μάλιστα ε, στα πλαίσια της ε, μακροπεριφερειακής στρατηγικής ε, του Ιουνίου ή της Αδριατικής Ιωνίου θάλασσας πειραματιστήκαμε σε μια καινούρια ιδέα ανάπτυξης τουριστικών δραστηριοτήτων με χώρες όπως η Αλβανία, όπως η Σερβία στο πλαίσιο αυτής της μακροπεριφερειακής στρατηγικής λοιπόν προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε επιχειρήσεις στο ιδιαίτερο πεδίο του πολιτισμικού τουρισμού, του πολιτιστικού τουρισμού. Είχαμε τρεις μήνες, 25 συμμετέχοντες, 11 testimonials που παρουσιάζονται σε όλη την Ευρώπη και 18 προτάσεις συγκεκριμένες ε, business plan που υπευλήθησαν. Οι θεματικές προφανώς έχουν να κάνουν με την πολιτική κληρονομιά της όλης αυτής μακροπεριφέρειας και επιχειρήσαμε να αναπτύξουμε σχέδια επιχειρηματικότητας για να βοηθήσουμε και τους σπουδαστές να παρακολουθήσουν αυτή τη διαδρομή και μετά μια αξιοποίηση, μια αξιολόγηση της ιδέας ε, με κριτικές προσεγγίσεις ε, ομαδικής εργασίας και άλλο ένα παράδειγμα και με αυτό θα κλείσω του πώς προσπαθήσαμε να αναπτύξουμε, να αξιοποιήσουμε ε, την μακροπεριφέρεια Αδριατικής Ιωνίου ήταν η δημιουργία του Ουνιάντριον που είναι ένα δίκτυο διαφορετικών πανεπιστημίων μισά ευρωπαϊκά και μισά από χώρε που δεν ειναι κρατήμελη αυτή τη στιγμή για να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα που διατίθενται από την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως το Erasmus Mundus και εδώ ενισχύουμε την κινητικότητα 184 σπουδαστών και ε, υποψηφίων διδακτόρων. Γιατί έτσι μπορούμε να δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες και δυνατότητες. Σας ε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ, λέει πρόεδρος, τον καθηγητή πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η παρουσίαση αυτής της μακροπεριφερειακής δραστηριότητας με, στα πλαίσια της οποίας ε, υπάρχει συνεργασία με τις υπόλοιπες βαλκανικές χώρες τα μη κρατημέλη και μια δικτύωση δηλαδή με διάφορους φορείς και σας ευχαριστώ που αναφερθήκατε και στην ε, διαφορετικότητα που είναι ένα από τα σημαντικά πλέον της Ευρώπης. Θα δώσω τώρα το λόγο στον ε, καθηγητή Σεφτσικ από το Πολυτεχνείο της Δρέσδης που θα μας μιλήσει για την ε, δημιουργία των ε, νεοσύστατων επιχειρήσεων. Παρακαλώ. Yes, thank you very much. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω για τον ρόλο των ε, πανεπιστημίων και των νεοσύστατων επιχειρήσεων στις ευρωπαϊκές στρατηγικές περιφερειακής καινοτομίας και θα σας δείξω σε 7 slide την κατάσταση στη Δρέσδη και τις συστάσεις που έχω για την ευρωπαϊκή πολιτική. Είμαι και και κοσμήτωρας ε, στο τμήμα επιχειρήσεων, αλλά είμαι και επικεφαλής της Επιτροπής για τη Δημιουργία Επιχειρήσεων, οπότε κοιτάζω αυτά τα θέματα σε καθημερινή βάση. Αν δείτε τη Σαξονία, είναι μια περιοχή όπου υπάρχει μια συγκεκριμένη στρατηγική καινοτομία ε, που έχει θεσπίσει η κυβέρνηση του κρατηδίου έτσι ώστε η κοινωνία, η οικονομία, η επιστήμη και οι άνθρωποι να συνδέονται σε μια ε, περιοχή που υπάρχουν λίγες μεγάλες επιχειρήσεις. Δεν μπορώ ε, να σας δώσω περισσότερες λεπτομέρειες γι' αυτό γιατί δεν έχω χρόνο, αλλά υπάρχει αντίστοιχη στο σελίδα διαδικασία αναδιάρθρωσης, παρόλο που υπάρχει πολύ χρόνος που έχει περάσει από την επανένωση των δύο Γερμανιών, η διαδικασία της αναδιάρθρωσης παραμένει ε, στο επίκεντρο. Προσπαθούμε να καλύψουμε το χαμένο ε, χρόνο. Είμαστε παρόλα αυτά πίσω από το μέσο όρο στη Γερμανία. Η οικονομία αποτελείται από μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις κάτι που δεν ισχύει μόνο στη Σαξονία, ε, σε όλη τη Γερμανία ισχύει, αλλά εμείς έχουμε ε, ένα, μια ιδιαίτερη εκπροσώπηση σε πολύ μικρές επιχειρήσεις. Οι μεγάλες που υπάρχουν είναι λίγες και έχουν έρθει εκεί λόγω δημόσιων επιδοτήσεων και έχουν περισσότερο εργοστάσια παρά τα κεντρικά, τα κεντρικά τους γραφεία. Στην Σαξονία έχουμε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα που είναι πάνω από το μέσο όρο. Αν δείτε τις στατιστικές, βλέπετε πόσες πατέντες δίνονται στη Γερμανία και σε αυτό το επίπεδο βλέπετε ότι η Σαξονία είναι από τις πρώτες περιφέρειες. Ε, έχει σηματοδοτηθεί η Σαξονία ως ε, μια αριστεύουσα περιφέρεια λόγω ακριβώς αυτού του πράγματος. Τώρα, η σχέση μεταξύ των νεοσύστατων επιχειρήσεων και των πανεπιστημίων. Είναι πολύ καλή η σχέση, είναι ένα πινκ-πονκ μεταξύ των δύο αυτών ε, κατηγοριών. Οι νεοσύστατες επιχειρήσεις οδηγούν στην καινοτομία τα πανεπιστήμια προχωρούν στην καινοτομία, αλλά δεν καλύπτουν το τελευταίο στάδιο, το πέρασμα στην αγορά. Όλα αυτά βέβαια ως αλληλεπίδραση είναι κάτι το θετικό. Οι startups φέρνουν την περιφέρεια και το πανεπιστήμιο σε νέους επιχειρηματικούς ε, τομείς. Ε, αυτό συνέβη και στη δική μας αλλά και σε άλλες περιφέρειες. Ας πούμε, δείτε πόλεις όπως το Dortmund πώς μεταμορφώθηκε. Για να δούμε ένα άλλο μέρος ε, της Γερμανίας. Αν δείτε τα νέα ταλέντα και πώς προσελκύονται, θα δείτε ότι στη Γερμανία ε, υπάρχουν πάρα πολλά ταλέντα στα πανεπιστήμια που παραμένουν για πολύ λίγο καιρό, εκτός από τους καθηγητές ενδεχομένως. Ε, και αυτό δεν έχει νόημα. Τα πανεπιστήμια προσπαθούν να αλληλοσυνδέσουν ε, τις ειδικότητε, ας πούμε οι μηχανικοί υπολογιστών ε, με άλλες ε, ειδικότητε προσπαθούν να φτιάξουν όλους τους κρίκους της αλυσίδας για να υπάρχει ένα ισχυρό μάρκετινγκ. Επίσης υπάρχει μια μεγάλη δεξαμενή ερευνητών που ιδάλλως δεν θα ήταν προσβάσιμη για την καινοτομία των επιχειρήσεων. Τουλάχιστον σε εμάς ε, δεν υπάρχει στη δική μας περιφέρεια μεγάλη έρευνα και καινοτομία εντός των επιχειρήσεων, εκτός αν είσαι μια μεγάλη αυτοκινητοβιομηχανία ή μια μεγάλη φαρμακευτική. Αν λοιπόν δεν υπάρχει αυτό σε επίπεδο εταιριών, αυτή η συνδυαστική κατάσταση είναι ιδιαίτερα σημαντική τι κάνουμε στο Πολυτεχνείο της Δρέσδης. Έχουμε μία ε, πρωτοβουλία υποστήριξη των πανεπιστημίων που συνδέει τα πανεπιστήμια και, τις και τα ερευνητικά κέντρα εκτός ε, Δρέσδης, εκτός πανεπιστημίου, ε, στην Δρέσδη και γύρω από τη Δρέσδη. Έχουμε 125 μάλλον έχουμε 20 με 25 startups κάθε χρόνο και πολύ ε, ε, περισσότερες, πολλά περισσότερα άλλα ωφέλη, όπως ας πούμε επιδοτήσεις για έρευνα. Αν έχει δημιουργηθεί ε, μία startup, για παράδειγμα, υπάρχει περαιτέρω δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ αυτής και των ερευνητικών κέντρων. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο συγχρηματοδοτεί αυτές τις πρωτοβουλίες, αλλά έχουμε και κονδύλια από την τοπική αυτοδιοίκηση, την περιφέρεια. Έχουμε τώρα τρεις κατηγορίες ε, ε, δράσεις. Πρώτον, πληροφόρηση και έβρεση ταλέντων. Προσπαθούμε να κλείσουμε το κενό, ε, το χάσμα στην πληροφόρηση που υπάρχει για το ευρύτερο κοινό. Στη Γερμανία ε, δεν υπάρχει πολλή γνώση σχετικά με το τι είναι η επιχειρηματικότητα. Άρα προσκαλούμε πολλές φορές ε, σημαντικούς επιχειρηματίες για να μιλήσουν σε 300-400 φοιτητές και άλλους ενδιαφερόμενους για να καταλάβουν πώς είναι ένας επιχειρηματίας. Επίσης βρίσκουμε ταλέντα, προσπαθούμε να έρθουμε σε επαφή με ερευνητές κάθε είδους και να αποκαλύψουμε πιθανές ιδέες και να τις προωθήσουμε περαιτέρω. Ο αριθμός των ιδεών που προσπαθούμε να προωθήσουμε είναι περίπου 70 με 80 το χρόνο. Κάνουμε μια ε, διαδικασία, έχουμε μια διαδικασία επιλογής, ένα φιλτράρισμα. Το επόμενο στάδιο και επίπεδο είναι η εκπαίδευση, όχι απαραίτητα ακαδημαϊκής φύσεως. Ε, μπορεί να έχουμε επιχειρηματική πρακτική εκπαίδευση για επιστήμονες κάθε είδους που κατά τα άλλα δεν θα είχαν δεξιότητες ε, για να φτιάξουν μια επιχείρηση ή άλλες προσωπικές δεξιότητες ε, και κοινωνικές δεξιότητες που χρειάζονται για να βρουν χρηματοδότηση για την startup. Επίσης έχουμε ομάδες που είναι κυρίως το ερευνητικό προσωπικό των πανεπιστημίων όμως έχουν περισσότερη λίγο εμπειρία από το μέσο όρο την ε, τοπική βιομηχανία. Προσπαθούμε λοιπόν μέσα από αυτούς να δημιουργήσουμε συνεργασίες ε, για να υπάρχει συμβουλευτική. Και στο τέλος έχουμε περίπου 20 με 25 startup το χρόνο. Οι μισές από αυτές είναι κυρίως στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας και συχνά προσπαθούν απεγνωσμένα να φτιάξουν την ομάδα τους. Και υπάρχει και το αντίθετο. Οι άνθρωποι με πολλές δεξιότητες προσπαθούν να πουλήσουν περισσότερο τις προσωπικές τους δεξιότητες. Όλα αυτά είναι πολλά υποσχόμενα. Έχουμε πολύ καλές startup στο επίπεδο της υψηλής τεχνολογίας, αλλά έχουμε και άλλες startups με χαμηλότερο προφίλ. Γενικά, έχουν δημιουργηθεί Πολλά ε, συνεργασίες μεταξύ των πανεπιστημίων και των ε, startups που διαρκούν στο χρόνο και ε, βοηθούμε τους πιθανούς ιδρυτές για να προετοιμαστούν. Τι θα μπορούσε να κάνει τώρα η ευρωπαϊκή πολιτική. Θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει μηχανισμούς όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, αλλά και άλλους τρόπους, όλα είναι ευπρόσδεκτα, για να επιτύχει δύο πράγματα. Πρώτον, να βοηθήσει τα πανεπιστήμια να κάνουν project σαν αυτά που περιέγραψα, αλλά και να βοηθήσουν τον κόσμο στα πανεπιστήμια να ανταλλάξει πρακτικές, ε, μεθόδους. Ανταλλαγή δηλαδή ε, όσο, ευρία, όσο περισσότερο ευρεία γίνεται. Είναι δύσκολο αυτές οι πρωτοβουλίες ε, να αυτοχρηματοδητηθούν και να προωθηθούν. Αυτό ήταν η νόρμα, η τυπική κατάσταση στη Γερμανία ως τώρα, αλλά δεν προχωρά. Θέλουμε επένδυση στις startups με οποιοδήποτε κερδοφόρο τρόπο, όχι μόνο επειδή δεν έχουμε τα εργαλεία για να επενδύσουμε σε αυτές τις startups. Οποιοςδήποτε γενικά επενδύσει πολύ νωρίς σε μία startup ε, τα τελευταία χρόνια δύσκολα θα, θα πρέπει να παλέψει για να έχει απο, απόδοση. Γιατί αυτό να αλλάζει στην περίπτωση των πανεπιστημίων. Γενικά μπορεί να παραπονιόμαστε για τα πανεπιστήμια. Ε, βλέπουμε ότι τα πανεπιστήμια έχουν ε, κατεύθυνση κυρίως προς τη δημιουργία γνώσης και έβρεση κοντιλίων και οι startups δεν έχουν κατά ανάγκη τέτοια προσέγγιση. Ίσως με την χρηματοδότηση θα μπορούσαμε να τους βοηθήσουμε με τις πρωτοβουλίες ανταλλαγής εκβέλτης των πρακτικών θα μπορούσαμε ας πούμε να αποφύγουμε την αναποτελεσματικότητα. Για παράδειγμα, ε, φαίνεται ότι πολλά πανεπιστήμια ε, πήραν μαθήματα από εμάς ε, σχετικά με το πώς να είναι αποτελεσματικές οι επενδύσεις σε τέτοια project. Ευχαριστούμε. Για την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η παρουσίαση και για την έκκληση που κάνατε να χρησιμοποιήσουμε περισσότερο και καλύτερα το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο που είναι πολύ ενδιαφέρουσα πηγή χρηματοδότησης για αυτές τις start-up. και να ασχοληθούμε πολύ πιο στενά με την ανάπτυξη της υπαίθρου, της ευρύτερης περιοχής όπου λειτουργεί το Πανεπιστήμιο. Τώρα, τελευταίος ομιλητής, κύριος Άλμπερτ Μπόιμερ, που είναι ηγετικός τέλεχος της CSB System και θα μας μιλήσει για την ανάπτυξη της υπαίθρου, της για την ε, συνεργασία μεταξύ του κόσμου επιχειρήσεων και της Υπέθρου. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θέλουμε λοιπόν μια συμβίωση μεταξύ Πανεπιστημίου και Υπέθρου. Είμαι ομιλητής από πλευράς της ΕΣΜΕ Ζουστέ Μαγκέ και είμαι υπεύθυνο για αυτήν την, ε, την εφαρμογή αυτού του προγράμματος. Πρώτα απ' όλα, δύο λόγια για την επιχείρησή μας για να καταλάβετε πώς συνεργαζόμεθα μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων. Είμαι Είμαστε στα σύνορα μεταξύ Ολλανδίας, Βελγίου και Γερμανίας και προσφέρουμε λύσεις ε, τεχνολογίας πληροφορής, ε, τηλεπικοινωνιών, λογισμικά δηλαδή, σε διάφορους τομείς, στην ε, φαρμακευτική βιομηχανία, τη χημική βιομηχανία και άλλους τομείς και τους δίνουμε και ε, λογισμικό και μηχανήματα και συμβουλές. Όλα αυτά τα κάνουμε ως μία επιχείρηση και η διαδικασία χορήγησης όλων αυτών συνδυάζεται. Τους δίνουμε και εκπαίδευση και υποστήριξη. Έχουμε πάνω από 20 γλώσσες ε, στις οποίες εργαζόμεθα και εκπροσωπούμεθα σε πάνω από 40 χώρες. Είμαστε διεθνής επιχείρηση και συνεργαζόμεθα με διάφορους άλλους που ασχολούνται με το τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας. Τα τελευταία χρόνια πήραμε διάφορα, διάφορες διακρίσεις. Θεωρείται πολύ καινοτόμο το ότι πήραμε μια διάκριση από το Ίδρυμα Bertelsmann ότι είμαστε, βοηθάμε τους ε, εργαζόμενους που θέλουν να έχουν και οικογένεια. Έχουμε λοιπόν κάθε δυνατότητα και για τους ε, πελάτες μας και για τους ε, εργαζόμενους μας και για όσους ενδιαφέρονται να συνεργαστούν μαζί μας. Στην περιοχή μας υπήρχε έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού και γι' αυτό αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε μία ανώτατη εκπαίδευση μαζί με το Πανεπιστήμιο του Ρήνου της Κολονίας. Αυτή η αντίληψη λοιπόν μας βοήθησε να αναπτύξουμε τις περιοχές της υπαίθρου και να ε, ε, αναπτύξουμε το επιστημονικό του δυναμικό. Έτσι βοηθούμε και τις επιχειρήσεις και όλη την ευρύτερη περιοχή και οι εκθέσεις του επιμελητηρίου της ε, Βόρειας Νανίας Βεσφαλίας δείχνουν που υπάρχουν ελλείψεις από πλευράς ειδικευμένου εργατικού δυναμικού. Εδώ στο χάρτη Βλέπετε τις αποστάσεις μεταξύ των διαφόρων ε, μεγάλων πόλεων Μένχεν Gladbach, Düsseldorf, Aachen, Köln. Αυτό είναι το αποφασιστικό κριτήριο για τους φοιτητές όταν αποφασίζουν πού θα σπουδάσουν. Πόσο κοστίζει, για παράδειγμα, η κατοικία, το αυτοκίνητο, το κόστος ζωής γενικότερα. Το Σεπτέμβριο πέρυσι μαζί με το Πανεπιστήμιο της ε, Κολονίας δημιουργήσαμε δύο ε, σπουδές πρώτα απ' όλα δίκηση επιχειρήσεων και ε, πληροφορική για τις επιχειρήσεις. Όλα αυτά είναι επιτυχημένα. Είναι φυσιολογικές σπουδές, 7 εξάμεινα bachelor και έχει και πρακτική εξάσκηση σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις. Δύο φορές ε, τη βδομάδα οι φοιτητές εργάζονται στο Πανεπιστήμιο και το Σάββατο. Πήραμε την αναγκαία διαπίστευση και αυτό αποδεικνύει ότι έχουμε επιτύχει πολλά αλλά έχουμε ήδη εργαστεί πολύ τα τελευταία χρόνια και ιδίως τους τελευταίους μήνες και τα προγράμματα σπουδών απευθύνονται σε άτομα τα οποία θέλουν, ενώ έχουν ήδη κάποιες σπουδές και ήδη εργάζονται, να αποκτήσουν περαιτέρω προσόντα. Τους τελευταίους μήνες φτιάξαμε τέσσερα νέα αμφιθέατρα και δαπανίσαμε 5 εκατομμύρια ευρώ. Είμαστε λοιπόν πολύ σημαντική επιχείρηση για τον τομέα της πληροφορικής στην περιοχή του Άχεν και θέλουμε να βοηθήσουμε τη μεταφορά γνώσης από τα πανεπιστήμια στις επιχειρήσεις. Στα νέα μας ε, αμφιθέατρα βλέπετε ότι υπάρχει η σωστή, ο σωστός εξοπλισμός και εργονομική διαρρύθμιση. Μέσω αυτού του νέου ε, κάμπους θεωρούμε ότι θα προσελκύσουμε περισσότερους φοιτητές που θέλουν να σπουδάσουν κοντά στο χώρο εργασίας τους και διαμονής τους. Η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Κολονίας είναι μια πολύ σωστή ε, συμβίωση μεταξύ ε, κόσμου των επιχειρήσεων και ε, των πανεπιστημίων. Χρησιμοποιούμε λοιπόν ήδη μόρφωση του μέλλοντος και εκπαίδευση του μέλλοντος ηλεκτρονικές μορφές ε, εκπαίδευσης κτλ. Είναι ιδιωτική η σχολή και αυτό σημαίνει ότι κάθε μήνα ε, ε, πληρώνουν δίδακτρα 360 ευρώ το μήνα. Αλλά το κόστος ενός διαμερίσματος στη Γερμανία είναι γύρω στα 350 ευρώ το μήνα. Δηλαδή είναι περίπου το κόστος ενός ενοικίου, το κόστος σπουδών. Ποιο είναι το όραμά μας για το 2020. Θέλουμε να έχουμε ένα αυτόνομο πρόγραμμα σπουδών για γενική διαχείριση επιχειρήσεων με τα κύρια κέντρα ε, προσοχής να είναι η βιομηχανία 4.0, ο προγραμματισμός για την επιχειρηματικότητα και οι φορητές σπουδές. Γιατί πρέπει να προσαρμοστούμε στις ανάγκες της αγοράς και γι' αυτό η επιχείρησή μας μέχρι το 2020 θέλει να απασχολεί γύρω στους 800 εργαζόμενους. Θέλουμε λοιπόν να υπάρξει ένα περιφερειακό πρόγραμμα ανάπτυξης για τους 15 για τους ανθρώπους 15 με 25 ετών που θέλουν να γίνουν προγραμματιστές λογισμικού. Έχουμε λοιπόν δημιουργήσει ένα είδος άδεια προγραμματιστή ως πιλωτικό πρόγραμμα. Θέλουμε να το εφαρμόσουμε τους επόμενους μήνες, καταρχάς στην περιφέρειά μας, αργότερα σε εθνικό και αργότερα σε ενωσιακό επίπεδο. Συμπέρασμα. Η καινοτομία στην εκπαίδευση δίνει φτερά στις περιφερειές. Ε, όποια επιχείρηση δεν ε, επενδύει στην κατάρτιση δεν έχει μέλλον. Γι' αυτό θέλουμε να το επιτύχουμε αυτό, για να αντιμετωπίσουμε τις νέες προκλήσεις και για τους εργαζόμενους και για τους ε, πελάτες μας και για ανθρώπους που θέλουν να σπουδάσουν από την περιοχή μας. Σε ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Πολύ ενδιαφέρουσα και αυτή η προοπτική, αυτή η παρουσίαση. Κάμερ Εύερτ, Μόργανο, ε, Γραμματικάκης. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ για τις τρεις πολύ ενδιαφέρουσες ε, παρουσιάσεις. Πολύ ενδιαφέρουσα η πρότασή σας κύριε Σεύτσικ. Αυτά δηλαδή που είπατε ότι δεν θέλουμε να προωθούμε μόνο την αριστεία αλλά πρέπει κατόπιν να μάθουμε στους νέους πώς να αξιοποιούν αυτές τις ιδέες. Για να φτιάξει μια επιχείρηση κανείς πρέπει να ξέρει πώς να έχει τα λογιστικά του σωστά, πώς να πληρώνει τους φόρους του. Όλα αυτά είναι θέματα που πρέπει να τα ξέρει. Δεν αρκεί η ιδέα. Άμα δεν ξέρει κανείς πώς να κάνει την ιδέα του επιχείρηση που να λειτουργεί, τότε κυριότερη startup πολύ σύντομα θα ταυτίσει. Και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ σωστή αυτή η παρατήρηση που κάνατε. Δεν είναι σημαντικό μόνο να έχουμε καλές ιδέες, αλλά κατόπιν να τις κάνουμε και επιχείρηση. Αυτή είναι η ερώτησή μου που απευθύνεται και στους άλλους. Υπάρχει συνεργασία, για παράδειγμα, με τους οργανισμούς για την ανάπτυξη της οικονομίας σε τοπικό επίπεδο, ούτως ώστε να βοηθούν τους νέους στη διαδικασία ίδρυσης επιχειρήσεων. Υπάρχει επίσης συνεργασία με τα επιμελητήρια για παράδειγμα. Δεν ξέρω αν στην Ιταλία αυτό το σύστημα επιμελητηρίων, εμπορικών, βιομηχανικών επιμελητηρίων. Θα ήταν όμως σημαντικό. Γιατί υπάρχει μια δυνατότητα ε, ε πολύ ευρύτερη συνεργασίας και αλληλοβοήθειας. Λοιπόν, ε, Μόργανο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τους εισηγητές τους για τις παρουσιάσεις τους. Εγώ σημείωσα τα εξή σημεία ως ερωτήσεις. Μου φαίνεται ότι για μία ακόμα φορά προκύπτει μια εικόνα κάπως υπερβολική που περιγράφει την Ευρωπαϊκή Ένωση διότι το θέμα είναι πώς μπορούμε να ανταγωνιστούμε σε διεθνές επίπεδο και επιτρέψτε μου να θυμίσω ότι η Κίνα μετά την έκθεση Σανγκάη έχει επενδύσει σε μεγάλο βαθμό σε μια σειρά εργαστηρίων έρευνας όπου οι προσωπικές επαφές διαματίζουν σημαντικό ρόλο. Ο πρώην πρόεδρος της Επιτροπής, ο κύριος Πρόντι, ε, μας θυμίζει ότι υπάρχουν χιλιόμετρα εργαστηρίων που δουλεύουν το ένα δίπλα στο άλλο. Εμείς έχουμε εξαιρετικά κέντρα ερεύνης, αλλά που δουλεύουν λίγο απομονωμένα. Το λέω αυτό γιατί και η επιχειρηματικότητα και η υποστήριξη των νεοσύστατων επιχειρήσεων ε, ε, ε, έχουν σχέση με τον πανεπιστημιακό χώρο. Δηλαδή η θεωρητική έρευνα τι σχέση έχει σήμερα με την εφαρμοσμένη έρευνα. Το λέω διότι αυτό έχει άμεση σχέση με τα πορίσματα, με τα αποτελέσματα που μπορούμε να έχουμε στον κόσμο της επιχειρηματικότητας και προκαλεί καθυστερήσεις. Και θα με ενδιαφέρει επίσης να καταλάβω ποια είναι η άποψή σας για την σχέση μεταξύ της ερευνητικής δραστηριότητας των πανεπιστημιακών φορέων και του περιεχομένου του διδακτικού. Και θα είχα και πολλά ακόμα να πω σχετικά με τις δημοσιεύσεις, τις ερευνητικές και άλλα. Και ίσως και εκεί θα άξιζε να παρατηρήσουμε κάποια πράγματα συγκρίνοντας με το διεθνές πλαίσιο που δεν μπορούμε παρά να συγκρινόμαστε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Λουίτζι. Ο κύριος Ματικάκης, παρακαλώ. Ε, θα είμαι πολύ σύντομος και πάλι τουλάχιστον έτσι ελπίζω. Ε, ο κύριο Λόγκη μου έκανε εντύπωση. Αναφέρατε δύο φορές, το σημείωσα, ότι για χίλιους κατοίκους υπάρχουν 100 startup, εταιρείε, επιχειρήσεις, κάτι τέτοιο. Δηλαδή κάθε οικογένεια είναι και μια, μια επιχείρηση περίπου αυτό. Ή δεν κατάλαβα καλά επιχείρηση. Τι είδους επιχειρήσεις είναι αυτές, ε, δηλαδή εντυπωσιακό. Και εγώ θα σας πρότεινα με όλη τη γνώση που έχετε ασφαλώς μια καλύτερη λέξη. Το contamination είναι αρνητικό. Υπάρχει η λέξη όσμωσης που είναι αρχαία ελληνική και αγγλική όμως σήμερα. Όσμωσης. Αυτό το πράγμα γίνεται. Αυτό είναι το παράδειγμά σας το οποίο ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ε, συζητήστε το λοιπόν εκεί μήπως και βαφτίσομαι απόψε ε, και επίσης ε, μου έκανε πολύ εντύπωση στην ομιλία του κυρίου Τσέσεκ. Γενικά πρέπει να πω κυρία Πρόεδρε προς τιμή σα και όσον την οργάνωσα ότι ο δεύτερος κύκλος επειδή πάει λίγο πιο πρακτικά ε, συμπληρώνει τον πρώτο και έτσι κάνει όλη τη σημερινή μερίδα εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Θα μπορούσαμε να μιλάμε επιμέρες Και εσείς μου έκανε εντύπωση υπήρχε μια αντιστοιχία start-up και κατά κάποιο τρόπο πανεπιστημίων. Δηλαδή είπατε και τη χαρακτηριστική λέξη σαν να υπάρχει πινκ-πονγκ, πράγματι, σαν να μην πέφτει ποτέ η μπάλα απ' έξω. Ε, σαν να μην υπάρχει φυλέ. Ε, πόσο καιρό έτσι χρονικά διαρκεί μια startup, πότε γίνεται επιχείρηση ή μονίμως μένει startup και παίζει πινκ-πονγκ με τα πανεπιστήμια. Ε, αυτά γενικά είναι ερωτήσεις, αλλά πραγματικά τίθενται τόσα θέματα που η απαντήσει είναι δύσκολες και εγώ το μόνο που λέω είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Ε. Ευχαριστούμε τον ε, Γιώργο. Η κυρία Τρούπελ παρακαλώ. Ευχαριστώ. Να απευθυνθώ στον κύριο Μπόιμερ. Ε, μας ε, περιγράψατε πολύ συγκεκριμένα την προσέγγιση σας σε πανεπιστημιακό επίπεδο και πραγματικά ήθελα να μάθω αν φτάνει να έχουμε πανεπιστήμια στις μεγάλες πόλεις. Ίσως να πάμε και στην περιφέρεια. Αυτό ε, στη δική σας περιφέρεια είναι κάτι που προβλέπετε, είναι κάτι σύνηθες, ε, τι γίνεται σε άλλες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με ενδιαφέρει, είναι αυτό η προσέγγισή σας ή προσπαθείτε να κάνετε αυτό που γίνεται σε άλλα μέρη. Μια τελευταία απάντηση, ε, ερώτηση πριν δώσετε απάντηση παρακαλώ. Ο συνάδελφος Λέκοφ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καλό απόγευμα σε όλους. Ε, Πολύ λυπάμαι που δεν άκουσα όλες τις παρουσιάσεις, αλλά με ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα. Εγώ προέρχομαι από την Επιτροπή Άγκρη, όπου συζητήσαμε την μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής και ένα, μία από τις θεματικές ήταν οι περιφέρειες και η ύπεθρος. Και στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν εξειδικευμένοι ηλεκτρονικοί μηχανικοί στην Βουλγαρία, συνήθως παραμένουν στα αστικά κέντρα Πώς μπορούμε λοιπόν να δημιουργήσουμε ένα σύνδεσμο μεταξύ της καινοτόμου επιχειρηματικής δραστηριότητας και της υπαίθρου, γιατί συνήθως η μεγάλη επιχειρηματική δραστηριότητα επικεντρώνεται στα αστικά κέντρα και η υπαίθρος χάνει το ανθρώπινο δυναμικό της, χάνει τους ε, εξειδικευμένους επιστήμονές της που πηγαίνουν να εργαστούν στις πόλεις. Πώς μπορούμε λοιπόν να υποστηρίξουμε τις δεξιότητες αυτές για να βοηθήσουμε της ε, περιφερεια. Υπέθρου. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Να προσθέσω τα εξή δύο, αν μου επιτρέπετε. Για τις δεξιο... την ανάπτυξη των δεξιοτήτων στην Ήπεθρο. Αυτή τη στιγμή έχουμε στη διάθεσή μας ε, ε, κάποια τμήματα πανεπιστημιακά ε, εξειδικευμένα για ακριβώς ε, την ανάπτυξη της υπαίθρου και βλέπετε ότι έχουμε ε, ελλείψεις, κενά εκεί, κάτι που θα μπορούσε να μεταφερθεί και στον κόσμο των επιχειρήσεων, αν θέλετε επαγγελματικά προφίλ. Πέραν δηλαδή της τεχνικής εκπαίδευσης που ήδη έχετε ενσωματωμένη στα πρόγραμμα, στο πρόγραμμά σας, ε, μήπως υπάρχει και κάτι προς αυτή την κατεύθυνση για να υποστηρίξουμε και την όσμωση που μας, μας προτείνει ο συνάδελφος Γραμματικάκης. Τώρα, για τα διπλώματα επίσης ευρεσιτεχνίας ήθελα να αναφερθώ. Γιατί έχουμε σημαντικές κοινοτομίες... οι οποίες μπορούν να είναι και, ε, ε, αν θέλετε, ένας παράγοντας ε, οικονομικής ε, ανάπτυξης, ε, οικονομικής δραστηριότητας και υπό την έννοια αυτή και προς την κατεύθυνση αυτή μπορούμε να κάνουμε κάτι περισσότερο γιατί από πλευράς των ερευνητών πολύ συχνά λέγεται ότι η υποβολή, η κατοχήρωση ενός διπλώματος ευρεσιτεχνίας έχει υψηλότερο κόστος και διερωτώ με αν θα μπορούσαμε και εμείς από πλευράς μας να κάνουμε κάτι για να βοηθήσουμε την προσπάθεια αυτή ώστε η έρευνα είτε η θεωρητική είτε η εφαρμοσμένη να μπορεί να έχει ένα πόρισμα, ένα αποτέλεσμα και ως ακαδημαϊκή δραστηριότητα και όχι ευρύτερα επιχειρηματική. Και αντίστροφα θα έλεγα να πάμε να ξεκινήσουμε από τον τελευταίο καθηγητή και να πάμε προς τον πρώτο. Κοιτάξτε, είμαστε σε μια περιοχή πέθρου Απέχουμε 30 χιλιόμετρα από το μεγαλύτερο αστικό κέντρο, από τον εγκύτρο αστικό κέντρο στη Γερμανία, λέμε μια παροιμία ανάλογη της Αθηνά και Χειρακίνη. Πρέπει όλοι να συνεργαστούμε και θεωρούμε ότι πρέπει να συνεργαστούν λοιπόν οι επιχειρήσεις, τα πανεπιστήμια και όσοι θέλουν να αποκτήσουν προσόντα. Έτσι λοιπόν ο επικεφαλής της επιχείρησής μας είπε να συνεργαστούμε με το Πανεπιστήμιο. Κατόπιν το Πανεπιστήμιο έδειξε πολύ καλή θέληση και δεν υπάρχουν πολλά παραδείγματα ε, όπου να πηγαίνουν οι επιχειρήσεις στα πανεπιστήμια. συνήθω γίνεται αντίστροφα. Αυτή τη μεταφορά της γνώσης μπορούμε να την διαμορφώσουμε. Το πανεπιστήμιο είναι πολύ ευέλικτο και εμείς κάνουμε έρευνα και είμαστε σε θέση να αποκτήσουμε και διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Πατέντες έχουμε 120. Έχουμε το δικό μας ε, ερευνητικό τμήμα όπως σας είπα. Παρ' όλα αυτά θέλουμε να κάνουμε περισσότερα για την εκπαίδευση στο εσωτερικό της επιχείρησής μας. Εργαζόμαστε και με άλλα πανεπιστήμια, στο Μόναχο, το Βερολίνο, τη Βόρεια Γερμανία και είμαστε διατεθειμένοι να συνεργαστούμε και με ξένα πανεπιστήμια. Ευχαριστώ πολύ. Να απαντήσω λίγες ε, ερωτήσεις για τις startup. Για τις startup μόνο μπορούμε να τις βοηθήσουμε στην αρχή. Μετά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Δεν μπορούμε να ε, παίζουμε το ρόλο συμβούλου ε, για τις επιχειρήσεις γιατί αυτό θα ήταν συναγωνισμός με τον κλάδο που χορηγεί συμβουλές όμως ε, οι επιχειρήσεις startup υψηλού επίπεδου πολύ σύντομα χειραφετούνται και φτιάχνουν δίκτυα συνεργάζονται μαξί τους άρα δεν ανησυχώ δεν μπορούμε να τους παράσχουμε δωρεάν συμβουλές αλλά συνεργαζόμαστε μαζί τους Τώρα για τα επιμελητήρια, τα εμπορικά επιμελητήρια. Βεβαίω, έχουμε στενέ σχέσει, συνεργαζόμαστε, δίνουν ε, επιδοτήσει στα άτομα πριν ξεκινήσουν τις νέες επιχειρήσεις και συνεργαζόμαστε. Υπάρχει δομημένη συνεργασία. Αλλά εμείς ως πανεπιστήμια και εκείνοι ω ε, επιμελητήρια έχουμε διαφορετικούς αποδέκτες. Εκείνοι ε, κυρίως προσπαθούν να βοηθήσουν ε, κανονικές επιχειρήσεις, συχνά μικρές, ενώ εμείς κυρίως ε, θέλουμε να βοηθήσουμε startup τεχνολογικού περιεχομένου. Εργαζόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον, γνωρίζουμε ένα τον άλλον, αλλά δεν παρεμβαίνουμε ο ένας ε, στο ρόλο του άλλου. Όσον αφορά τις δημοσιεύσεις, εμείς δίνουμε, συγγνώμη, την βοήθεια γενικότερα. Δεν δίνουμε απευθείας χρηματοδότηση από τους πόρους της έδρα μου, για παράδειγμα, για τα startup. Δεν μπορώ να χρηματοδοτήσω startup. Όμως στη Γερμανία έχουμε αυτή την ιδέα του Humboldt ότι η έρευνα και η διδασκαλία πρέπει να συνδέονται. Βοηθάμε επιχειρήσεις ε, να αποκτήσουν πρόσβαση σε επιχειρηματικό κεφάλαιο. Εμείς στην έδρα μου το κάνουμε, γιατί κάνουμε έρευνα για τον τρόπο απόκτηση επιχειρηματική ε, χρηματοδότησης, επιχειρηματικού κεφαλαίου. Και έχουμε κάνει καλή έρευνα σε αυτό το τομέα και τα απορίσματά τη ακριβώ μας βοηθούν να δώσουμε συμβουλές στις επιχειρήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ ο κύριος Λόγγε, ο καθηγητής Ευχαριστώ. Είναι πολλές οι ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλες. Έχουμε ένα δίκτυο του εμπορικού επιμελητηρίου που επεκτείνεται σε όλη τη χώρα στην Ιταλία ε, και εντός αυτής της δομής συνεργάζονται όλες αυτές οι δραστηριότητες ε, επιχειρηματικότητας ε, που αποτελείται από ενώσεις, ε, φορείς, ε, οργανισμούς, επιχειρήσεις, τράπεζες που χρηματοδοτούν αυτού του είδους τη δραστηριότητα. Είναι σαφές ότι <clears throat> εμείς δεν μπορούμε να έχουμε αρμοδιότητα επί εργαστηρίων σε εκατοντάδες χιλιόμετρα συνεχούς γραμμής όπω είπε ο συνάδελφο, αλλά μπορούμε να αξιοποιούμε τα αποτελέσματα της δουλειά των εργαστηρίων. Αυτή είναι η πρόκληση που έχουμε μπροστά μας. Δηλαδή, έχουμε σημαντικά κονδύλια, σημαντικούς πόρους, ε, σημαντική τεχνολογία. Δεν μπορούμε παρά να αξιοποιήσουμε τη δουλειά τους. Ε, μιλώ, ας φέρω ένα παράδειγμα πρακτικό. Η διάχυση των smartphones ή των κινητών τηλεφώνων αυτό βασίζεται στην τεχνολογία, αλλά όχι μόνο. Η διάχυσή τους βασίζεται στην εξή απλή ιδέα. Της προπληρωμένης κάρτας SIM. Δηλαδή, το μέσο με το οποίο ε, προβαίνουμε σε, μια, σε ένα συμβόλαιο χωρίς να υπάρχει συμβόλαιο, αν θέλετε να το πούμε έτσι. Από εκεί πέρα ήρθαν και οι τεχνολογικές λύσεις, αλλά η κεντρική ιδέα που ήταν η επιτυχής ιδέα ήταν η ιδέα της παροχής μιας υπηρεσίας υπηρεσία για την οποία υπήρχε ανάγκη. Επ' αυτού πρέπει να εργαστούμε, να συνεργαστούμε με όσμωση, όπως είπε ο κ. Γαματικάκης, Ναι, υπάρχουν διάφορες ειδικεύσει και αρμοδιότητες που συνεισφέρουν. Απλώς ε, εμείς σκεφτήκαμε και γλωσσικά, αν θέλετε, αυτήν την ιδέα της ε, contamination ε, ως κινητήριο μοχλό αυτή της δραστηριότητας αλλά εν πάση περιπτώσει το σημαντικό είναι ε, το ποσοστό της συμμετοχής των ε, νεοσύστατων επιχειρήσεων στην Ιταλία. Εγώ είχα την ευκαιρία να το παρουσιάσω αυτό. Και το μεγάλο ποσοστό που συμμετέχει στα πανεπιστήμια. Στη δική μας περιφέρεια όλα αυτά είναι δομημένα γύρω από την Πανεπιστήμια της Αγκώνα. Στο βορρά είναι γύρω από το Πανεπιστήμιο του Τρέντο. Επομένως υπάρχει αυτός ο ρόλος των πανεπιστημιακών φορέων ο καταλητικός. Γιατί ακριβώς υπάρχει η πρώτη υπάρχει η ιδέα, υπάρχει η προσπάθεια. Ίσως ποσοτικά να μην ε, έχουμε τα ιδανικά αποτελέσματα, αλλά ποιοτικά οπωσδήποτε είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που συμβαίνει. Και έχουμε καινούργιε ιδέες. Από εκεί και πέρα ε, αυτό θα πρέπει να γίνει σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα της έρευνας γιατί όλη μας η σταδιοδρομία σε αυτό βασίζεται, στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της ε, έρευνας. Αν υπήρχε η δυνατότητα λοιπόν εισαγωγή και μιας αξιολόγησης της βοήθειας που παρέχουμε στην ε, επιχειρηματικότητα μεταξύ των νέων, είναι για παράδειγμα μία παράμετρος που μπορεί και αυτό να ενσωματωθεί στους δείκτες αξιολόγησης. Χρειαζόμαστε αυτή την κινητήριο δύναμη που θα οδηγήσει σε ανάπτυξη. Ανάπτυξη οικονομική για τι και, και οι μικρές επιχειρήσεις τι οποίες αναφερθήκαμε νωρίτερα είναι ένα, μια μέση αξία, ένα μέσο μέγεθος. Υπάρχουν και πολύ μικρές και πολύ μεγάλες. Αλλά μεταξύ του συνόλου των επιχειρήσεων στην περιφέρεια ε, έχουμε μικροεπιχειρήσεις οι οποίες παράγουν ε, αυτήν την παραγωγή υψηλής ποιότητας υποδημάτων, προϊόντα design ιταλικού για παράδειγμα, όπου η τοπική τεχνογνωσία αριστεία ε, καθιστά τη δραστηριότητα αυτή υψηλά ανταγωνιστική. Αυτό είναι ένα πρότυπο διακεχημένο στην Ιταλία. Αλλά είναι και πρόβλημα γιατί έχουμε να κάνουμε με πολύ μικρές επιχειρήσεις. Διότι ο συνδυασμό των μικρών επιχειρήσεων με τα εργαστήρια δεν είναι πολύ εύκολο. και χρειάζεται λοιπόν ομαδοποίηση αυτή τη προσπάθεια. χρειάζεται μια δομή, μια αρχιτεκτονική, ένα οικοσύστημα που θα επιτρέψει σε όλες αυτέ τις διαφορετικές μικρές επιχειρήσεις να αναπτύξουν τη δυνατότητά τους την ανταγωνιστική. Και μάλιστα όχι μόνο σε περιφερειακό αλλά σε διεθνές επίπεδο. Αυτή είναι η πρόκληση της παγκοσμιοποίησης και στην περιφερεια μα. Και την πρόκληση αυτή εμείς την αποδεχθήκαμε, την αναγνωρίσαμε, ώστε να αναγνωρίσουμε αγορές, δυνατότητες στην αγορά και δυνατότητες συνεργασίας και παραγωγικής συνεργασίας. Επομένως, το σκεπτικό είναι ότι από την διαφορετικότητα μπορούν να, δημιουργηθεί, να δημιουργηθούν δυνατότητες. Επίσης έχουμε απομακρυσμένες περιοχές της Πέθρου και ορεινές περιοχές στην Ιταλία. Έχουμε τα απένινα που διασχίζουν όλο το μήκος της χώρας ε, και τα πρόσφατα ήταν ε, συζητήθηκαν πολύ λόγω του σεισμού, αλλά έχουμε αραιοκατοικημένες περιοχές ορεινές, οι οποίες όμως θα μπορούσαν επίσης να είναι δυνατότητα ανάπτυξης οικονομικής για αυτές τις περιφέρειες. Εδώ μας χρειαζόμαστε πολιτικές, ευρωπαϊκές αλλά και εθνικές, που θα είναι σε θέση, που θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν όλη αυτή τη διαφορετικότητα. Γιατί και σε αυτά τα οικοσυστήματα υπάρχει υψηλότατη ποιότητα ζωής. Ε, και μέσω της διαφορετικότητας αυτής μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτές τις περιοχές αντί να τις θεωρούμε απομακρυσμένες ζώνες της υπαίθρου. Ευχαριστούμε, λέει η Πρόεδρος, για αυτήν την παθιασμένη συνεισφορά, θα έλεγα. Εγώ θα κλείσω λέγοντας το εξής. Εμείς με μεγάλη χαρά και ενδιαφέρον σας ακούσαμε, συζητήσαμε μαζί σας, είχα ζητήσει και από την γραμματέα ε, να συλλέξει όλες αυτές τις πολύτιμες παρουσιάσεις ε, για να μπορέσουμε να τις ε, διανύμουμε όχι μόνο στους συναδέλφους Επιτροπής αλλά και στους συναδέλφους άλλων επιτροπών και ίσως να την ανεβάσουμε και στην ιστοσελίδα μας. Και ήθελα να συνοψίσω λέγοντας τα εξή. Πρώτον, εμείς παρακολουθούμε προσεκτικά και είμαστε διαθέσιμοι να μας θεωρήσετε τακτικούς συνομιλητές πέραν αυτής της σημερινή συζήτησης γιατί αυτή την περίοδο μαζί με την Επιτροπή Εργασίας εξετάζουμε το σύνολο του θεματολογίου των δεξιοτήτων θεωρούμε ότι εσείς μπορείτε να συνεισφέρετε με πολύτιμο τρόπο σε αυτό. Υπάρχει η επερχόμενη ανακοίνωση της Κομισιόν για την, τον εξυγχρονισμό των ανώτων δομών εκπαίδευσης, όπως μας είπαν οι πρόσωποι της Κομισιόν, και αυτό είναι θέμα που μας ενδιαφέρει να συζητήσουμε μαζί σας και ίσως θα σας ζητήσουμε και συνεισφορές συγκεκριμένες και νομίζω ότι και στην εφαρμογή των προγραμμάτων του Ορίζοντα, του Erasmus Plus και άλλων θα θέλαμε πραγματικά να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να υλοποιήσουμε τους στόχους μια ε, πληρέστερη συμμετοχή των πανεπιστημιακών φορέων, όχι μόνο στην κινητικότητα των σπουδαστών, αλλά και σε άλλες δράσεις ε, πολύ σημαντικές κεντρικής σημασίας, εταιρικών σχέσεων, ε, διδακτικών συστημάτων και με τη συμμετοχή των κεντρικών πανεπιστημίων. Νομίζω ότι σήμερα είδαμε με σαφήνεια πόσο ενδιαφέρουσα είναι μια τέτοια συζήτηση ε, για την τρίτη αποστολή, όπως έλεγα, των πανεπιστημίων, δηλαδή ε, ως φορέων όχι από, μόνο, όχι από μόνους τους, ε, φορέων όμως που μπορούν να οδηγήσουν στην οικονομική ανάπτυξη. Νομίζω ότι η, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προσέξει αυτόν τον νέο ρόλο, τον ενισχυμένο ρόλο που μπορούν να αναλάβουν τα πανεπιστήμια και να δοθούν προσδοκίες ε, κατεύθυνση στη νέα γενιά, στη νεολαία, δυνατότητα σύσταση νέων επιχειρήσεων, νέου πνεύματος επιχειρηματικότητας. Νομίζω ότι η εμπειρία της δικτύωση είναι πολύ σημαντική σε αυτό το πλαίσιο, όχι μόνο στην διαδικασία της Μπολόνια, αλλά στα διάφορα δίκτυα και σε επίπεδο μακροπεριφερειών που υπάρχουν. Και κλείνοντα ε, θα αναφερθώ λίγο στο ranking. Όταν η Επιτρόπος Βασιλείου πρόσφατα ε, πρότεινε αυτή την αξιολόγηση, τη βαθμολόγηση των πανεπιστημίων και όλοι ξέρουμε ε, το ευαίσθητο του θέματος, εν πάση πτώση ήταν ένα σύστημα ranking. Ο βαθμός διεθνούς παρουσίας θα έπρεπε να λαμβάνεται υπόψη, λέμε εμείς. Η επίτροπο λέει ότι πρόκειται για ένα μεταβατικό κριτήριο που είναι η δυνατότητα ανάπτυξης επιχειρηματικότητας. Νομίζω ότι και αυτό είναι ένα στοιχείο που θα μπορούσαμε να ενσωματώσουμε και να το υποβάλουμε ως πρόταση στην ε, Γενική Διεύθυνση. Πάντως είναι σημαντικό να μην χάσουμε τις παρουσιάσεις σας. Θα έχουμε λοιπόν ε, μια ε, συνοπτική παρουσίαση των παρεμβάσεών σας και σας ευχόμαστε πολύ καλή δουλειά γιατί τη χρειαζόμαστε τη δουλειά σας. Ευχαριστούμε. Eh, eh, ε, να πω το εξή. Θα θυμάστε ότι αύριο στις 3.30 το απόγευμα Έχουμε την επίσκεψη στην ΕΑΤΣΕΑ, ε, στον Οργανισμό Εκπαίδευσης. Αύριο λοιπόν στις 3.30 και την Πέμπτη έχουμε την ψηφοφορία για την έκθεση για το EICC. Για, τις, ε, για τη βιομηχανία, την πολιτιστική και τη δημιουργική. Ευχαριστώ.